Okay. Um, λοιπόν, καλημέρα. Ξέρετε ότι είχαμε αναβάλει την ψηφοφορία και γι' αυτό έχουμε περισσότερο χρόνο. Είμαστε στο 7 τώρα, εκλογή αντιπροέδρου. Και θα δώσω πρώτα το λόγο στην Ελίσσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη γλώσσα του Σέξπιρ για να τα πω πιο γρήγορα. Η νέα συνάδελφος Ματλεν Μιζή είναι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής ήταν όταν, από τότε που έφυγε ο Εδουάρδος Σικλούνα. Προτείνω λοιπόν να πάρει τη θέση του επίσημα ως πλήρες μέλος και να το δεχτεί επίσημα η Επιτροπή. Μήπως θέλει κανείς να αντιμιλήσει ή μπορούμε να συμφωνήσουμε διαβοή. Διαβοής. Ναι. Ελάτε λοιπόν τώρα εδώ επάνω για να καταλάβετε τη θέση σας. Και ένας από τους, α ναι, μπράβο, ευχαριστώ. Είναι σαν να ανεβαίνετε τη σκάλα στις κάνες, ορίστε. Λοιπόν, σαμπάνια δεν έχουμε σαμπάνια, ούτε καν αφρόδι γιατί κάνει οικονομίες στο Κοινοβούλιο Λιτότητα. Για να δούμε τώρα λοιπόν αν συγκρατηθείτε τη ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης. Είναι πάντα περίεργο όταν προεδρεύω για δική μου γνωμοδότηση, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι το εννέα. Ας μην κάνουμε ενδεικτική ψηφοφορία. Θα δούμε αν υπάρχουν όλες οι κάρτες όταν φτάσουμε εκεί λοιπόν. Τροπολογία 1 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 2 τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβατή τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται νομίζω τώρα όμως πρέπει να επαληθεύσουμε με τις κάρτες Λοιπόν ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 5 5 Άρχισε η ψηφοφορία, αλλά πρέπει να προσθέσουμε και μια ψήφο για μένα. Λοιπόν, ψήφισατε όλοι με ακόμα ένα. Έληξε η ψηφοφορία. Καλά αυτό ακυρώνουν, αλλήλο ακυρώνονται. Λοιπόν έληξε η ψηφοφορία, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά θα το ξαναεπαληθεύσω. με τις ομάδες θα απορριπτόταν, όμως θα εγκρινόταν, αλλά με τις παρουσίες μπορεί και να απορριφθεί. Λοιπόν, και ένας παραπάνω υπέρ λοιπόν, μετρήστε, απορρίπτεται. Οχτώ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται Παρά αυτά που λέει το χαρτί, περνάμε τώρα στη συμβιβαστική Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στο δεύτερο τμήμα νομίζω εγκρίναμε κάτι που δεν είναι λογικό τέλο 16 με προφορική τροποποίηση. Μήπως έχει κανείς αντίρρηση για την προφορική τροποποίηση. Όχι. Μάλιστα. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά το σύνολο όπως έχει τροποποιηθεί και μία ψήφωση παραπάνω υπέρ. 37 υπέρ, μία ψήφος κατά, τρεις αποχές. Ευχαριστώ. Είχαμε πει ότι θα δούμε τι θα κάνουμε για τον φόρο. Αλλά μετά από συζητήσεις φαίνεται ότι η συγκήτρια τώρα είναι διατεθειμένη να αναβλεβάλει την ψηφοφορία μέχρι τις 17-18 Ιουνίου ελπίζοντας να έχει επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τότε. Ζήτησε μία συμφωνία υπό όρους για να φτάσουμε τον Ιούλιο στην Ολομέλεια, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε τέτοιους όρους. Ούτως ή άλλως η διάσκεψη των Προέδρων θα καθορίσει τι πάει και τι δεν πάει στην Ολομέλεια. Εγώ θα έλεγα ότι θα αναβάλουμε την ψηφοφορία μέχρι τότε ελπίζουμε να επιτευχθεί πρόοδος και αν δεν επιτευχθεί τότε θα πρέπει να το ξαναδούμε. Ελπίζω ότι οι ομάδες θα καταφέρουν να συμφωνήσουν. Μπορεί να χρειαστεί να το επαναπέμψουμε στην Επιτροπή. Αν φανεί ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, δεν μπορούμε να πάμε στην Ολομέλεια. Η Άννη ζήτησε το λόγο. Θέλεις πρώτος εσύ ούντο. Όχι η Άννη. Και αν χρειαστεί μπορούμε να ψηφίσουμε και τώρα. Ίσως αυτό να κάνουμε γιατί όπως είπαμε χθες είχαμε πει ότι αν χρειαστεί θα το κάνουμε. Ιάννη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, είπατε και εσείς, ε, καταλήξαμε σε μια συμφωνία να αναβάλουμε τη ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ μέχρι τις 17 Ιουνίου και αυτό μας δίνει κάποιο περιθώριο ελιγμών για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η συζήτηση για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών έχει διαρκέσει τα τελευταία τρία χρόνια. Έτσι λοιπόν είναι απόλυτα εφικτό να καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι τις 17 για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Απλώς ήθελα να τονίσω ότι αυτός ο στόχος να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ούτε έχει ζητήσει το λόγο. Πρόεδρε. Ε, εγώ Άκουσα τι είπατε εσείς ε, για τις ε, ψηφοφορίες χωρίς όρους, ε, όμως εγώ ξέρω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιείται αυτή η λύση για να πάει το ζήτημα στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Πάντως, εγώ σέβομαι αυτό που είπατε, προέδρε, ότι πρέπει να υπάρχει διακριτική ευχέρεια και το να οριστεί μια ημερομηνία ψηφοφορία είναι για να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου. Πρόεδρος, ναι. Αλλά όπως σας είπα, η ημερομηνία δεν είναι κάτι που εξαρτάται μόνο από τους εισηγητές. Ο Μάρκους, με ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επιδεινώνουμε τα πράγματα. Ξέρουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν συζητήσει αυτό το θέμα και συμφωνώ με την πρόταση της εισηγήτριας εδώ. Θέλω να συμβάλλω και εγώ για να μπει αυτό στην ημερησία διάταξη, στην ε, διάσκεψη των Προέδρων και κατόπιν στην Ολομέλεια. Γιατί να κάνουμε τα πράγματα πιο δύσκολα όπως είναι στην πραγματικότητα. Πρόεδρος, μάλιστα, αυτό που προτείνω είναι να αναβάλουμε την ψηφοφορία μέχρι τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 17-18 Ιουνίου Ελπίζουμε τότε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή και αν συναντήσουμε δυσκολίες μπορούμε να το ξαναδούμε. Αλλά ο στόχος αυτή τη στιγμή θα ήταν να ψηφίσουμε σε εκείνο το στάδιο και υπάρχει χρόνος για να πάμε και στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Αν αποτύχουμε, αν δεν τα καταφέρουμε, τότε θα το ξαναδούμε. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Ο Επιτροπός Αλμούνια λογικά θα έπρεπε να έρθει στις 10.30. Επομένως, σας κάνουμε 10 λεπτά διάλειμμα μέχρι να φτάσει ο Επίτροπος. Εντάξει, ευχαριστώ.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 Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Αλμούνια εδώ στη συνεδρίασή μας. Πάντοτε είναι πρόθυμος να έρχεται. Συνήθως εμείς είμαστε που έχουμε το πρόβλημα να βρούμε αρκετό χρόνο για να συνομιλήσουμε μαζί του, αλλά χαίρομαι που παρευρίσκεται εδώ σήμερα. Θα ακολουθήσουμε τη συνήθη διαδικασία ανταλλαγή απόψεων Καταρχήν, θα ακούσουμε τον Επίτροπο και κατόπιν θα έχουμε ερωταπαντήσεις ε, σε χρόνους 5 ε, λεπτών. Έχετε 10 λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ την Επιτροπή ΕΚΟΝ και την Πρόεδρο που μου δίνει και πάλι την ευκαιρία να παρευρεθώ ενώπιόν σας και να σας παρουσιάσω την ετήσια κρίση ανταγωνισμού για το 2012. Πέρσι συνεχίσαμε να εργαζόμαστε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον για την επιβολή της νομοθεσίας ε, σχεδόν 6 ε, χρόνια από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ευρώπη προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις βαθιές ε, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες από όσα αναδύθηκαν και συνέβησαν το 2007 και το 2008 και πάλι είναι περισσότερο επιτακτικό από ποτέ να εφαρμόσουμε την πολιτική ανταγωνισμού την Ευρωπαϊκή Ένωση με εύρωστο τρόπο και επίσης να μιλήσουμε για την συγχώνευση και τον έλεγχο, των αντιτράστ και τις κρατικές ενισχύσεις. Ε, μαζί με το κανονιστικό έργο της Κομισιόν αντιγηθήκαμε σε χαμηλές ε, ε, τιμές για τους καταναλωτές και για επιλογή όταν χρειάζομαι. Επίσης ενδυναμώθηκε η ενιαία αγορά βάσει των δρασεών μας και βλέπουμε κάποιους τομείς που λειτουργούν στα πλαίσια της μοντέρνας οικονομίας όπως το χάρη πάρει, τις ενεργειακές, ε, ενεργειακούς τομείς, τηλεπικοινωνίες ε, και ε, πέρσι επίσης δείξαμε την αποφασιστικότητά μας να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη ε, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Και το Μάιο ξεκίνησαμε τη στρατηγική του εξυγχρονισμού της κρατική, των κρατικών ενισχύσεων και θα σας ενημερώσω σχετικά επίσης. Θα παρουσιάσουμε ε, επίσημα μια πρωτοβουλία για την ιδιωτική επιβολή του νόμου επιβλή στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, πέρσι αρχίσαμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τις τράπεζες που βρίσκονται σε δυσκολίες με στόχο ένα πιο διαφανή χρηματοπιστωτικό τομέα. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης θα μας παρέχει μας παράσχει το πλαίσιο που χρειαζόμαστε για να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας. Μεταξύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο είναι κοντά στην εθέτηση της νέας νομοθεσίας για την εξυγίανση των ε, τραπεζών. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα να διασφαλίσουμε τη μετάβαση ε, προς ένα νέο υγιές κράτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο να θεωρούμε τους κανόνες κρατικής ενίσχυσης για να συνάδουν με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αναδυθεί σε σχέση με τη δράση μας πέρσι αναλάβαμε, λάβαμε 19 αποφάσεις ε, και αυτή η δική κανόνας κρατικών ενισχύσεων για το χρηματοπιστωτικό τομέα μεταξύ αυτών από τότε που ξεκίνησε αυτό το πλαίσιο κρίσης έχουμε λάβει 62 αποφάσεις ε, και ε, αποφάσεις ε, ανοικοδόμησης και ρευστοποίησης και έχουμε τώρα κάποιες εκκρεμείς υποθέσεις πάνω από 20. Να υπενθυμίσω την διάρθρωση του τραπεζικού τομέα στην Ισπανία. Ήταν ειδικέ αυτέ οι αποφάσει γιατί ελήφθησαν βάση μνημονίου συνεννόηση που υπεγράφει τον Ιούλιο, πέρσι τον Ιούλιο. Όλε οι σχετικέ αποφάσει ε, ε, ε, δύο, γερμανικά, δύο γερμανικές τραπεζές, μία από τη Λετωνία και τη δεξιά Επίσης χρησιμοποιήσαμε και μέσα σε άλλες περιπτώσεις. Θα θυμάστε ότι η πιο σχετική απόφαση πέρσι ήταν η απαγόρευση της συγχώνευσης μεταξύ της, ε, του Euronext ε, και του χρηματιστηρίου της Γερμανίας. Επίσης, συνεχίσουμε το έργο μας ε, για τις εταιρείε πιστοτικών καρτών. Επίσης ξεκινήσαμε μία έρευνα για να ερευνήσουμε κάποιες πτυχέ της δράσης της Mastercard και πριν δύο εβδομάδε η Visa Europe ε, προσέφερε να μειώσει ε, τα τέλη για τις πιστοτικέ κάρτες και να διευκολύνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πέρσι η Κομισιόν συνέχισε το έργο της για δύο έρευνε αντιτράστ που ξεκίνησαν το 2011 ε, την αγορά των credit default swaps ε, και επίσης ε, τα ε, ποσοστά benchmark που αφορούσαν μια σειρά τραπεζών και διαμεσολαβητών. Επίσης κάναμε κάποιους ελέγχους σε καταστάσεις τραπεζών αλλά και στον τομέα των βιοκαυσίμων και Επίσης, ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν έχουν κάνει σιωπηλή συμφωνία για τη χειραγώγηση των τιμών οι εταιρείε. Μια άλλη σημαντική περίπτωση στον τομέα τη ενέργεια αφορά την Gazprom. Ξεκινήσαμε επίσημε διαδικασίε αντιτράστ πέρσι. Επίση, η δράση μα στο ενεργειακό τομέα συνάδει με τον ε, κανονιστική δουλειά που γίνεται στα θεσμικά όργανα. Η δημιουργία μια αυθεντική ενία ε, αγορά ενέργεια για του χρόνου έχει επανεπιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περισμένης εβδομάδας. Επίσης, αναπτύξαμε και την νομοθεσία ενιαίας αγοράς και στις τηλεπικοινωνίες πέρσι. Είχαμε μια περίπτωση με την Τελεφώνικα και την Τέλεκομ της Πορτογαλίας και ε, λάβαμε κάποιες ε, αποφάσεις ε, που αφορούσαν τον ανταγωνιστική εταιρεία Orange και επίσης Πέρσι ε, φέραμε την πρώτη νέα γενιά, ε, την επικοινωνιών μέσα στο πλαίσιο ξεχρονισμού θέλουμε να έχουμε ανταγωνιστικές και καινοτόμες αγορές ε, στις ψηφιακές βιομηχανίες. Επομένως, θέλω να τονίσω δύο αποφάσεις που λάβαμε πέρσι και μία περίπτωση που εκκρεμεί στις αποφάσεις μας για τα ηλεκτρονικά βιβλία δεχτήκαμε τις δεσμεύσεις της Apple ε, και τεσσάρων ε, εκδοτών στην μουσική βιομηχανία που ε, είναι ένα μεγάλο τμήμα της ψηφιακής βιομηχανίας. Συμφωνήσαμε με τη Universal και την EMI αφού λάβαμε σημαντικές παραχωρήσεις και τέλος έχουμε την συνεχιζόμενη περίπτωση antitrust με την Google. Αυτή είναι μια επισκόπηση των κυρίων φυχών. Ε, των δράσεων επιβολής του νόμου πέρσι, το Μάιο του 2012, η Κομισιόν ξεκίνησε την ε, θέση σε εφαρμογή της στρατηγική εξυγχρονισμού κρατικών ενισχύσεων. Αναπτύσσεται πλήρως αυτή η διαδικασία. Θα έχουμε και τις ε, νέες κατηγορίες γραμμές για την περιφερειακή βοήθεια που θα υιοθετηθούν τον επόμενο μήνα και θα διευκολύνουν την εφαρμογή κάποιων κανονισμών. Την περσμένη εβδομάδα διθέτησε σχετική έκθεση και επιτροπή, επιτροπή Έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια για το περιβάλλον, για το κεφάλαιο κινδύνου και προβλέπεται και η οθέτηση κανονισμού σχετικά με τη ξενολόγηση του κινδύνου ε, για το επόμενο εξάμενο ή αρχές του 2014. Ελπίζω ότι η στρατηγική εξυγχρονισμού στο σύνολό της ε, θα έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τα μέσα του 2014. Επίσης, θέλω να αναφέρω την πρωτοβουλία του Antitrust και την διαδικασία ελέγχου των συγχωνεύσεων και θα ε, παρουσιάσω την πρόταση για το Antitrust στους συναδέλφους την επόμενη εβδομάδα για το 2011 τη σχετική έκθεση ανταγωνισμού θα την παρουσιάσω προς η θέτηση δυνάμει της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας. Ε, θα είναι η πρώτη φορά στον τομέα του ανταγωνισμού που θα γίνει κάτι τέτοιο και θα σας παρουσιάσω τα κύρια χαρακτηριστικά των προτάσεών μας αμέσως ε, μετά την έγκριση από την Κομισιόν. Ελπίζω ότι με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτής της Επιτροπής θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε ταχαίως την πρόταση. Όταν το πράξουμε θα έχουμε πετύχει δύο στόχους κοινού. Καταρχήν να διευκολύνουν ε, τις μεγάλες ε, ομάδες ε, παραβίασης του νόμου να λάβουν την κατάλληλη αποζημίωση και δεύτερον να υπάρξει παρκής εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα του. Επίσης θα κάνουμε πιο φιλικές προς τη χρήστη της αξιολογήσεις των διάφορων περιπτώσεων, θα θετήσουμε μία πλουστευμένη διαδικασία για να, ή, για μειωθεί η ποσότητα των πληροφοριών που παρέχουν οι εταιρείε σε μη προβληματικές περιπτώσεις, θα επιταχυνθεί η διαδικασία και θα επικεντρωθούμε σε πιο προβληματικές συγχωνεύσεις. Παράλληλα, σκεφτόμαστε αν ο έλεγχος των συγχωνεύσεων θα πρέπει να επιτεθεί και στην απόκτηση ε, των ε, μετόχων ε, που δεν ε, ανήκουν στη μειοψηφία, γιατί σήμερα έχουμε δει κάποια προβλήματα και δεν έχουμε μέσα να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά ίσω θα χρειαστεί να τροποποιήσουμε τον κανονισμό συγχωνεύσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρξει μια δημοσία διαβούλευση για αυτό το θέμα του επόμενου μήνε. Εμεί ε, εξετάζουμε ένα σύστημα παραπομπής ε, που θα, ε, εξε... όπου θα εξετάζονται οι περιπτώσει μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών. Και θέλω να αναφερθώ και στη συνεργασία μα με άλλου οργανισμούς πριν να ολοκληρώσω πέρσι η Κομισιόν συνέχισε να συνεργάζεται με τις αρχές υπηρεσίες ανταγωνισμού εντός ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού για να ενθαρρύνει ε, τη σύγκληση και να εφαρμοστούν ομοιόμορφα οι κανόνες αντιτράστ. Πρέπει να αναφέρω ότι η συνεργασία αυξάνεται με τις εθνικές αρχές. Το τελευταίο παράδειγμα είναι η συμφωνία που υπογράφει πριν λίγες ημέρες με την Ελβετική ε, πλευρά και θα εγκριθεί και από το Ελβετικό Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά η Κομισιόν θα μπορεί να ανταλλάξει αποδεικτικά στοιχεία με μια αρχή ανταγωνισμού τρίτης χώρας χωρίς ε, να ε, υπάρχει ειδική εξαίρεση για την εταιρεία. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολλά μπορούμε να κάνουμε για την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση και για να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάκαμψη, πρέπει να συνεχίσουμε να μειώσουμε τα επίπεδα του χρέους για καλύτερη κατανομή των προσπαθειών και των θεσιών, πρέπει να υποστηρίξουμε την κατάρτιση, την έρευνα, την κοινοτομία. Και Επίσης πρέπει να ολοκληρώσουμε το project της Τραπεζικής Ένωσης και να εμείνουμε στις προσπαθίες μας για να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η ενιαία αγορά. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι σημαντική συνιστόσα σε αυτό το μείγμα πολιτικής, γιατί μέσω της επιβολή της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς, να βελτιώσουμε το επιχειρησιακό περιβάλλον και να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη. Ξέρω ότι είναι κοινή αυτή η στόχη και αυτό το όραμα και θέλουμε να πετύχουμε όλα αυτά μαζί σας μέσω του διαλόγου και ιδίω μέσω της σχέσης μας με την ομάδα ανταγωνισμού που δημιουργήθηκε από εσάς. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα θα περάσουμε στις ερωτήσεις, στις ερωτοπαντήσεις, να ζητήσω από τους βουλευτές να προσπαθήσουν να μην υπερβούν τα δύο λεπτά γιατί αν υπερβείτε το χρονικό όριο των δύο λεπτών θα πρέπει να σας σταματήσω. Δεν μπορούμε να έχουμε τόση ώρα. Για το ΕΛΚ ο κύριος Γκοζέζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εδώ είμαι εδώ. εδώ. Με χάσατε, όχι έψαχνα την Ισπανική καμπίνα λοιπόν. Σας ευχαριστώ για την προσέλευση σας. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όλα όσα είπατε. Αλλά επιτρέψτε μου να θέσω ένα ερώτημα που μπορεί να σας φαίνεται ασήμαντο, αλλά που παρόλα αυτά ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις και την αντίληψη που έχουν οι πολίτες για να καταπολεμηθεί η κλοπή και κατακράτηση μετάλλων η Γαλλία θέλησε να διευθετήσει την πώληση σιδηρούχων μεταλλευμάτων που ξέρετε ότι κλέβουν σύρματα που περιέχουν ε, χαλκό και τα ξαναπουλάνε. Και γι' αυτό ο νόμος της 6ης Ιουλίου 11 απαγορεύει την ε, πληρωμή της μετρητής σε ιδιώτες ορισμένων μετάλλων, σιδηρούχων και μη. Υπάρχει όμως εδώ το αναπάντεχο αποτέλεσμα ότι δεν το κάνουν το ίδιο και άλλες χώρες μέλη και άλλα οι περιοχές κοντά στα σύνορα συνεχίζουν να σημειώνουν ε, τέτοιες παράνομες πωλήσει ή κλοπές με στόχο να πουληθούν στη γειτονική χώρα. Γι' αυτό το πολύ ασήμαντο λοιπόν θέμα η Κομισιόν προβλέπει καμία εναρμόνιση. Έχει τεθεί το ερώτημα και στη Γαλλική Βουλή και ο Υπουργός είπε ότι θα έπρεπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει κάτι έτσι ώστε η καταπολέμηση να είναι αποτελεσματική σε ολόκληρη την Ένωση. Σας επαναλαμβάνω μπορεί να μην είναι πολύ σημαντικό θέμα αλλά είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς βλέπουν οι πολίτες την Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Γκοζέσου. Δεν μπορώ όμως να σας απαντήσω γιατί το θέμα αυτό όσο σημαντικό και να είναι είναι θέμα του συμπατριώτη σας Μιχαήλ Μπαρνιέ. Oui, si vous permettez, Ναι, αλλά ε, όταν σκέφτεται κανείς τον ανταγωνισμό, εσάς σκέφτεται. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θέλω να υπησέλθω στα θέματα των συναδέλφων μου. Υπάρχει ένα σχετικό θέμα εδώ πέρα, ξαναλαβαίνετε, σε ό,τι αφορά τη χρήση των αγαθών ως ε, εγγύησης και κατά πόσο θα μπορούσαμε με τον τρόπο αυτό να αποφύγουμε ένα ε, ενδεχόμενα μονοπόλια. Θα το συζητήσω αυτό ίσως και αργότερα και ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε τα, τις πρώτες δηλαδή ως ενδεχόμενη εγγύηση και πώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πώς ε, ε, οδηγεί σε έλλειψη των υλών αυτών. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες σκέψεις, ίσως και σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για τα benchmarks. Να περάσουμε στους σοσιαλδημοκράτες. Η Ελίζα Φερέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ που παρευρίσκεστε εδώ. Έχω δύο ερωτήσεις και οι δύο σχετικές με την Τραπεζική Ένωση και συγκεκριμένα με την νέα οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών και την δημιουργία της Αρχής Εξυγίανσης και του Ταμείου Εξυγίανσης. Μία τράπεζα ως δομή που βασίζεται σε καταθέσεις και με μικρό ενεργητικό πέρα από τις καταθέσεις για να μπορεί να γίνει διάσωση με μέσα στην περίπτωση εξυγίανσης θα ε, θέσει περισσότερο σε κίνδυνο τους καταθέτες από μια πιο πολύπλοκη τράπεζα η οποία θα έχει πιο πολλά στρώματα πάνω από τους καταθέτες αυτό θα σημαίνει ότι οι πιο υγιείς τράπεζες, δηλαδή αυτές που βασίζονται πιο πολύ σε καταθέσεις, θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερο για να διασφαλίσουν αυτές οι ίδιες καταθέσεις από τις πιο πολύπλοκες και πιο αδιαφανείς τράπεζες που de facto στην πρακτική τελικά ε, τους εγκαιώται μία περισσότερη πιθανότητα να διαφυλάξουν τις καταθέσεις. Έτσι λοιπόν οι πιο ε, σίγουρες τράπεζες ε, θα έπρεπε να αντισταθμίσουν τον κινδύνο προσφεύγοντας περισσότερο στις καταθέσεις. Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης και θα ήθελα να ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε για το ζήτημα αυτό. Το δεύτερο ερώτημα, πολύ σαφές είναι το εξή. Η νέα νομοθεσία για την επίλυση των κρίσεων δεν εμποδίζει να συνεχίζει να γίνεται το bailout των τραπεζών, η διάσωση των τραπεζών. Έτσι λοιπόν πώς η ε, πολιτική ανταγωνισμού θα εγγυηθεί ότι πιο ισχυρές οι χώρες δεν θα συνεχίσουν να κάνουν bailout τραπεζών, δηλαδή να διασώζουν τις τράπεζες ε, με χρήματα των φορολογουμένων, ενώ οι τράπεζες που βρίσκονται σε πιο αδύναμες χώρες θα πρέπει να προβαίνουν στο μπέιλινγκ, in στη με διαμέσα και επομένω θα πλήττονται και οι καταθέτες ε, και οι μέτοχοι και οι πιστωτές. Έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και είναι ακριβώ το αντίθετο που, στο οποίο, με αυτό στο οποίο αποσκοπεί η Τραπεζική Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φερέιρα. Το πρώτο σημείο στο οποίο αναφερθήκατε εσείς δεν είναι ακριβώς ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να επιληθεί από μέσω των αλληλεγγύων των κρατικών ενισχύσεων. Εγώ με τη δική σας ανησυχία, είναι αλήθεια πως ε, αν ε, μια τραπεζική οντότητα δεν έχει στο εισήγειό της επαρκές κεφάλαιο μέσω των, δράσ, μέσω των μετοχών, επαρκεί μέσα για να απορροφήσει τις απώλειες ε, ή ε, χρέη τότε φτάνουμε στον ε, κατάλογο αυτό που λένε ε, οι Άγγλοι Pecknotter και φτάνουμε τότε στο στο χρέο, στο senior debt ή στις καταθέσεις που ε, εκεί έχουμε τις καταθέσεις αυτές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, άνω των 100.000 δηλαδή και κάτω των 100.000 που καλύπτονται από την εγγύηση. Υπάρχει υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ε, τραπεζών που έχουν μια σχέση μεταξύ του ενεργητικού τους και των καταθέσεών τους πολύ ισορροπημένη και υπάρχουν συγκριτικά τράπεζες που έχουν μία δομή στο παθητικό τους που να εξαρτάται πολύ περισσότερο από την πρόσβαση στην αγορά και εξαρτάται λιγότερο από τους καταθέτες. Αυτό δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων, όπως είδαμε και στην περίπτωση της Κύπρου. Μπορούμε κάτι τέτοιο να το δούμε, ίσως ε, οριακά και στο μέλλον, σε περίπτωση εξυγένσης άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων. Εγώ συμμερίζομαι την ανησυχία σας, αλλά από τη σκοπιά του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων πρέπει να διευκρινίσω πώς όλα όσα σημαίνουν ε, ε, συνεισφορά του ήδη, της ίδιας της τράπεζας να χρηματοδοτήσει το κόστος της εξηγίασής της δεν ε, μπαίνει ως θέμα κρατικών ενισχύσεων εξορισμού. Οι κρατικές ενισχύσεις επισέρχονται από τη στιγμή που το Ίδρυμα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την εξηγίασή του με, ίδιους φόρους και πρέπει να προσφύγει σε δημόσια κονδύλια ε, ή σε κάποιους πόρους όπου εισέρχεται εκεί και η κρατική ενίσχυση. Έτσι λοιπόν, περισσότερο είναι ένα θέμα Συμβουλίου Κοινοβουλίου που αυτή τη στιγμή συζητούν την οδηγία της ε, ανάκτησης και εξυγίανσης παρά ένα θέμα που μπορεί να επιληθεί από τη σκοπιά των κρατικών ενισχύσεων. Τώρα, όταν μπαίνει το θέμα των κρατικών ενισχύσεων είναι στη δεύτερη περίπτωση που, στην οποία σας αναφερθήκατε που συνδέεται με την πρώτη. Όταν ε, μπαίνει ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων σε μία διαδικασία εξυγίανσης, γίνεται αυτό όταν χρησιμοποιούνται πόροι δυνάμει των κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή εθνικοί πόροι στα ταμείου εξυγίανσης είναι κρατική ενίσχυση. Χρηματοδοτούνται, είτε χρηματοδοτούνται από την τράπεζα, είτε μεικτός από την τράπεζα και από το δημόσιο τομέα. Δεν έχει σημασία. Ένα ταμείο εξυγένση είναι κρατική ενίσχυση, ένα εθνικό ταμείο εγγύηση καταθέσεων επίση είναι κρατική ενίσχυση και η χρήση των χρημάτων οικονομικών πόρων ε, του μηχανισμού ESM είναι επίσης κρατική ενίσχυση. Αν στο μέλλον υπάρχει ένα ταμείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα κοινό ταμείο εξυγίανσης ε, με αμοιβαιοποίηση δεν θα είναι κρατική ενίσχυση. Όμως το βαθμό που το Ταμείο δεν ε, είναι αμοιβαιοποιημένο για το σύνολο των κρατών μελών είναι κρατική ενίσχυση. Και κάθε φορά που υπάρχει προσφυγή σε τέτοια ταμεία μπαίνει το θέμα του έλεγχου των κρατικών ενισχύσεων. Τι προετοιμάζουμε τώρα για να αφαιρήσουμε το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο του ελέγχου κρατικών ενισχύσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Κάποιε νέε κατευθυντήριε γραμμέ που ελπίζω να μπορέσουν να εγκριθούν πριν από το καλοκαίρι, όπου δυνάμει τη εμπειρία που έχουμε και κυρίως στην ισπανική περίπτωση και τις απόφαση που ελήφθη από την Ολλανδική κυβέρνηση με αυτό το πραγματικό SNS. Δηλαδή, να μην θεωρείται συμβατή η ενίσχυση κρατική όταν προσφεύγουν σε ταμεία δημόσια αν πριν δεν είχε γίνει το bail-in σε τρία επίπεδα. Τα τρία πρώτα επίπεδα του καταλόγου προτίμησης. Μέτοχοι, κάτοχοι βρυδικών προϊόντων με δυνατότητα απορρόφησης απολειών και δευτερεύων χρέων. Πιστεύουμε ότι η χρήση δημοσίων πόρων θα πρέπει να προηγείται μιας διαδικασίας ε, μάλλον θα πρέπει να ακολουθεί αυτή τα τρία στάδια του Μπέιλιν της διάσωσης μέσα. Δεν πάμε παραπέρα. Σε. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό και αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα επικάλυψης σε ό,τι αφορά τα κονδύλια για την υποστήριξη των τραπεζών, των καταθετών και της ε, κρατικής ε, επένδυσης μέχρι ε, ότου συλλέξουμε και χρήματα από τον κλάδο αυτό. Αυτό είναι το μήνυμα και είναι μάλλον αρκετά περίπλοκο. Ο Ραμών από την Άλτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα θα μιλήσω τη γλώσσα του κυρίου Ελμούνια. Γιατί διάβαζα τα απομνημονεύματα του Ζαν Μονέ και ε, παρουσιάστηκαν στα καταλανικά. Έτσι λοιπόν θα σας ε, μιλήσω στη γλώσσα σας. Λέω, ο Επίτροπος, αν μπορείτε να μιλήσετε καταλανικά, εγώ σας καταλαβαίνω. Ελπίζω μια μέρα να είναι δυνατόν όλα θα γίνουν. Αν εσείς ε, το 2000 είχατε κερδίσει τις εκλογές, ίσως ε, να μην ε, ήμασταν στη σημερινή κατάσταση. Αλλά ας φτάσουμε στα θέματα που μας αφαιρενόζαν. Μονέ, τι θα μας έλεγε. Θα μας έλεγε πως ε, η τραπεζική πίστοση σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλη για την οικονομική αναπτύξη, όπως ήταν σημαντικός ο άνθρακας και στη δεκαετία του 50 και σε όσους βρισκόμαστε εδώ σήμερα ίσως ε, θα μας έλεγε να επικεντρωθούμε στην ε, σταθεροποίηση στην παγίωση της Τραπεζικής Ένωσης πριν από τις ευρωεκλογέ, πριν από οτιδήποτε άλλο. Να επικεντρωθούμε δηλαδή στο να αντιμετωπίσουμε τον κατακαιρματισμό ε, της τραπεζικής πίστοσης. Γιατί στην περίπτωση που μας απασχολεί, οι χώρες του Νότου κάθε φορά έχουμε πρέπει να πληρώνουμε όλο ένα και περισσότερα για το δανεισμό, ενώ σημαίνει ακριβώς το αντίθετο στις βόρειες χώρες. Έτσι, λοιπόν, θέλω να ρωτήσω σε ποιο βαθμό στην Ισπανία έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για την εξυγίανση των τραπεζών, αλλά ε, παρόλα αυτά δεν υπάρχει ροή αυτής ε, της ε, πίστοσης, παρά την προσπάθεια λοιπόν εξυγένσης του τροπεζικού τομέα. Οι τρεις μεγάλες τράπεζες στην Ισπανία θα έχουν τα τρία τέταρτα των μεδίων της αγοράς. Πιστεύετε ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ της μείωσης διαθέσιμης πίστοσης με την αύξηση της συγκέντρωσης. Δεν θα ήταν δυνατό να συνδέσουμε τις κρατικές ενισχύσεις με το να υπάρξει πίστοση στην οικονομία. Ευχαριστώ κύριε Τρεμόσα, ο κύριο Σαλμούνια. Εγώ συμφωνώ μαζί σας στο ότι είναι επίγον να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν και να ολοκληρώσουμε με το πιο αξιόπιστο τρόπο την Τραπεζική Ένωση. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι επίγον και είναι και απαραίτητο. Δεν λέω πως, ε, και, πως δεν έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα και συζητήσεις ε, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στον οικονομικό τομέα, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στο δημοσιονομικό τομέα, σε βιομηχανικούς τομείς, για την ενέργεια, για τις τηλεπικοινωνίες. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Όμως, αυτή τη στιγμή η πίστοση είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, χωρί πίστοση. Πολύ δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε πώ μπορούμε να πετύχουμε σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή στρατηγική. Οτιδήποτε και γίνει σε άλλου τομεί ή με άλλε πολιτικέ. Στην περίπτωση τη Ισπανία. Εγώ δεν πιστεύω πως ε, είναι πολύ λογικό ή ότι θα είναι αποτελεσματικό το να σκεφτούμε ότι η πίστοση θα προέλθει από τις τράπεζες που έχουν περισσότερα προβλήματα στην Ισπανία. Κυρίως όταν σκέφτομαι το πόσο ε, χρειάζεται να αυξηθεί η πίστοση στη μη χρηματοπιστική οικονομία. Εμείς ε, είδαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν δημόσιοι πόροι, αλλά παρόλα αυτά ε, συνέχιστηκαν να υπάρχουν δυσκολίες στην περίοδο της κρίσης. Όμως ε, πολλές ε, φορές έγινε εξηγήση των προϋπολογισμών, υπήρξε πρόσβαση στην αγορά. Εγώ νομίζω ότι οι τράπεζες που... Οι τράπεζες είναι αυτές που θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσουν ε, τις πιστοτικές ροές. Τώρα πώς θα το κάνουν αυτό, η εντύπωσή μου είναι ότι πρέπει να δούμε την πλευρά της ζήτησης, της πίστοσης και αυτό ε, σχετίζεται με πάρα πολλούς ε, παράγοντες, με την ύφεση και με κάποιες ε, πολύ εύθραστες οικονομικές προσδοκίες, βραχυπρόθεσμα, όμως πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα για αυτό το τομέα, γιατί η πολιτική πρέπει να εξυπηρετεί όλη την οικονομία, όχι μόνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στα πλαίσια του χρηματοπιστωτικού συστήματο κάναμε μια ενίσχυση των συζυγίων των τραπεζών, για την εξυγίαση των τραπεζών και αυτέ οι προσπάθειε ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίαση των υγιών τραπεζών ε, δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τις πιστοτικές ροές που χρειάζεται η οικονομία. Στην Ισπανία έχουμε προβλήματα τώρα και στη ζήτηση και στην προσφορά τη πίστοση. Όμω για την προσφορά τη πίστοση δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει επανενεργοποίηση, ιδίω από τι τράπεζε που είναι τώρα σε διαδικασία αναδιάρθρωση. Απαραίτητη μεν, αλλά πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζητάμε από αυτέ να κάνουν περισσότερα από ό,τι κάνουν άλλε τράπεζε. Και είναι αλήθεια ότι το επίπεδο τη συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα στην Ισπανία αυξήθηκε λόγω των συγχωνεύσεων, επειδή εξαφανίστηκαν κάποια και οντότητες, όμως αν συγκρίνουμε την ισπανική αγορά με άλλες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι το πιο συγκεντρωμένο σύστημα το ισπανικό. Νομίζω ότι έχει μια δομή σε ό,τι αφορά το ρόλο και τον αριθμό των οντοτήτων που επιτρέπει υγιή ανταγωνισμό μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Thank you. το κουμπί. Ο Ζαν Πολμπέση από τους Πράσινους, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Καλώς ορίσατε. Μας κάνατε έναν απολογισμό της, του προγράμματος της Κομισιόν για τον ανταγωνισμό. Πολύ εξαντλητικό. Υπάρχει όμως ένα θέμα που για μας έλειπε και που είναι μάλλον στρατηγικό για μας τουλάχιστον ανώ ένα ψήφισμα της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής του Ιανουαρίου 13 για τον εξυγχρονισμό της πολιτικής dans son 6 στο θέμα των κρατικών χρεών και έλεγε ότι η πολιτική του ανταγωνισμού πρέπει να επιτρέπει τις δημόσιες ενισχύσεις, τις κατάλληλες δημόσιες ενισχύσεις για, την οικολογική, για τον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας με περισσότερη χρήση ανανεωσίμων και περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας. Και ότι αυτό λέει θα έπρεπε να είναι η βάση των νέων καθευθυντηρίων γραμμών της πολιτικής ανταγωνισμού. Για μας δεν είναι ασήμαντο και δευτερεύον θέμα έτσι διακοσμητικό, αλλά μία πιθανή δυνατή βάση της μελλοντικής πολιτικής και δραστηριότητας και απασχόλησης και δημιουργίας πλούτου μπροστά στην αναγκαιότητα εξοικονόμησης των πόρων. Ερωτώ λοιπόν αυτό το θέμα που για μας έχει στρατηγική σημασία τι απέγινε στο πρόγραμμά σας. Το κριτήριο αυτό συμπεριλαμβάνεται στη γενική σύλληψη του ανταγωνισμού που έχει η Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Μπέσερ. Ευχαριστώ κύριε Μπέσερ. Προηγουμένως είχα πει έτσι συνοπτικά ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που θα ενημερωθούν πριν λήξει η θητεία σας και μίλησα για την ενέργεια και το περιβάλλον. Μέχρι τώρα οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν το περιβάλλον μόνο, αλλά αυτή τη φορά, γιατί αυτό μας δείχνει η εμπειρία, πρέπει να το συνδυάσουμε και με την ενέργεια. Και γι' αυτό προετοιμάζουμε τώρα κάνουμε τις πρώτες δημόσιες διαβουλεύσεις και συζητήσεις μία από τις κατευθύνες γραμμές θα είναι και ενέργεια περιβάλλον μαζί και βέβαια μεταξύ των νέων αυτών γραμμών θα αφιερώσουμε σημαντικό τμήμα στις ανανεώσιμες ενέργειες που πρέπει να την χάνουν δημόσια στήριξη, ήδη την χάνουν, να θα συνεχίσουν μέσω της χρήσης όχι μόνο των προκαθορισμένων στόχων από την Ένωση αλλά ήδη και για μετά το 2020 αλλά λοιπόν και με βάση την, τα συμπεράσματα από τα εθνικά προγράμματα στήριξης της ανανεώσιμες ενέργειες που η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού αναλύει αυτή τη στιγμή. Μελετάει. Θα συνεχίσουμε φυσικά να στηρίζουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι απολύτως απαραίτητο. Και μπορούμε ήδη να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα από την εμπειρία των περασμένων ετών. Καμιά φορά μερικές ανανεώσιμες πηγές θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ανταγωνιστικές χωρίς δημόσια στήριξη. Αυτό είναι πολύ καλό νέο, ότι ας πούμε η ολική ενέργεια, υπό ορισμένες συνθήκες βέβαια, μπορεί να είναι ανταγωνιστική χωρίς δημόσια στήριξη που είχε μέχρι τώρα. Και το άλλο στοιχείο είναι, για να μην μακρηγορήσω τώρα, ότι τα αποκλειστικά εθνικά προγράμματα στήριξης της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να είναι μεν απαραίτητα γιατί δεν υπάρχει αρκετή διασύνδεση πανενωσιακός και γι' αυτό η ενιαία αγορά ενέργειας είναι και αυτή ένας προ... στόχος πρωτεύων αλλά η συγκέντρωση των στηρίξεων σε εθνικές μονοπροσπάθειες καταλήγει σε κάποιο κατακαιρματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς ενεργείας και οι εθνικές επιλογές δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τις επιλογές των γειτονικών κρατών και άρα η χρησιμοποίηση δημοσίων στηρίξεων για τις ανανεώσιμες πηγές πρέπει να έχει μια ευρωπαϊκή πτυχή διάσταση. Αλλιώς, ενώ συμμεριζόμαστε όλοι το στόχο, θα καταλήξουμε σε κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς. Και τώρα από το ECR. Thank you. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το ερώτημα που έχω να σας θέσω είναι απλό και εύκολο αν θέλετε και μάλιστα το θίξατε το θέμα αυτό εν συντομία κατά τις ε, εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Πριν από δύο εβδομάδες η Επιτροπή ξεκίνησε χωρίς ε, ευθυνδιαστικές επιθεωρήσεις κάποιων ενεργειακών ε, εταιριών και μια εταιρεία που σε ό,τι αφορά τις ε, αναφορές αυτές. Αν προκύψει ότι οι εταιρείε αυτές όντως είχαν ε, χειραγωγήσει τις τιμές ε, των, της ενέργειας σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την παροχή αερίου. Η ζημιά προς τους καταναλωτές ήταν τεράστια και ρωτώ λοιπόν τι θα συμβεί αν η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμα στις εταιρείες αυτές για παραβίαση των κανόνων κατά της σχηματισμού μονοπωλίων. Και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανταποκριθεί στις αξιώσεις των ε, καταναλωτών που θα προκύψουν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τρέτσεκ. Όπως είπατε, πριν από κάποιες εβδομάδες, πριν από δύο εβδομάδες συγκεκριμένα νομίζω, κάναμε ευθυνδιαστικές επιθεωρήσεις σε κάποιες ε, πετρελαιό ε, βιομηχανίες ε, και σε κάποιες πλατφόρμες. Αναφερθήκατε στις πλάτς. Και λάβαμε εκθέσεις από τις εταιρείες αυτές για ορισμό benchmark σε ό,τι αφορά τις τιμές του πετρελαίου και για άλλες τιμές ενέργειας. Σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα αυτό μοιάζει κάπως με τα benchmark στον ε, χρηματοοικονομικό κλάδο και στις ερεύνες που διεξάγουμε και σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες ε, ε, νοθείες, σε ό,τι αφορά τον ορισμό των benchmarks, σε ό,τι αφορά την χρήση των εκθέσεων, σε ό,τι αφορά τον ορισμό των benchmarks που ανακοινώνεται κάθε ημέρα στους ε, φορείς της αγοράς. Και παράλληλα μπορεί να υπάρχει ε, παραβίαση των νόμων του ανταγωνισμού που ενδεχομένως να δίνει όφελος σε αυτούς που κάνουν την ε, εσφαλμένη, τον εσφαλμένο ορισμό των τιμών. Σε περίπτωση που λοιπόν διαπιστωθεί τέτοια παραβίαση, αυτό φυσικά δεν μπορούμε να το προκαταλάβουμε, γιατί βρισκόμαστε σε φάση ε, διεξαγωγής ακόμα των επιθεωρήσεων, θα ε, ληφθεί απόφαση για επίσημη έρευνα σε ό,τι αφορά τον, τα χρηματοοικονομικά benchmarks. Ερευνούμε και παραβιάσεις βάσει του νόμου κατά τον καρτέλ και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 101 και 102 άρθρα της συνθήκης. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω όμως τι θα γίνει με τον τομέα τον ενεργειακό αν ακολουθήσουμε το διπλό αυτό δρόμο του άρθρων 101 και 102 ή αν θα χρησιμοποιήσουμε ένα από τα δύο αυτά άρθρα σε ό,τι αφορά τις συνέπειες σε περίπτωση που έγινε όντως τέτοια παραβίαση και τέτοια παραποίηση, αν διαπιστωθεί αυτή η παραποίηση, όντως στην περίπτωση αυτή θα είναι τεράστιες οι ζημιές οι οποίες έχουν υποστεί οι καταναλωτές και οι χρήστες. Από πλευράς πολιτικής ανταγωνισμού, αναφέρθηκα και εισαγωγικά σε αυτό, σε κάποιες εβδομάδες θα υποβάλουμε μια πρωτοβουλία νομοθετική για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που θα επιτρέψει να ζητήσουμε αποζημίωση από τις, ε, σε ό,τι αφορά ζημιές που προκλήθηκαν από παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την νομοθετική μας ε, πρωτοβουλία προκειμένου να εγκριθεί με συναπόφαση το συντομότερο δυνατόν. Κάποια κάτι μέλη προβλέπουν σχετική εθνική νομοθεσία, αλλά χρειαζόμαστε και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Όπως ξέρετε, το Κοινοβούλιο συζήτησε τα θέματα αυτά στη σχετική έκθεση που ψηφίστηκε πλειοψηφικά στην Ολομέλεια. Θέματα συλλογικών αγωγών. Θα πρέπει να περάσουν από πιο πολλή έρευνα προτού μεταφραστούν σε νομοθεσία σε, ε, ό,τι αφορά ε, αποζημίωση για περιπτώσεις παραβιάσεων της, ε, του νόμου περί ανταγωνισμού. Και θα λάβατε αυτή την ε, νομοθετική πρωτοβουλία το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Κλούτα από την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Κύριε Επίτροπε, δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Καταρχάς, υπάρχει μια αντιπαράθεση με την εταιρεία Google υπήρξαν προβλήματα, συγκεκριμένα η Google. Οι πελάτες της Google που είχαν χρησιμοποιήσει τις ε, διαφημίσεις της και είχαν έτσι καλύτερη και υψηλότερη θέση σε περιπτώσεις αναζήτησης μέσω της Google. Είχαν προβλήματα σε σχέση και με τους ε, άλλους πελάτες της Google. Ε, έγιναν λοιπόν κάποιες ερωτήσεις, μια έρευνα, λάβαμε μια απάντηση από την Google η οποία δεν είναι πολύ ικανοποιητική σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτή. Ποια είναι η στάση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δεύτερη ερώτηση που κινείται προς τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Το έδειξα και στην προηγούμενη συνάντησή μας σε ό,τι αφορά τους γαλακτοπαραγωγούς. Ε, ήρθαν εδώ στα τέλη του προηγούμενου έτους και στην αρχή του τρέχοντος έτους και μας ε, έχησαν πάρα πολύ γάλα. Έκαναν μια σχετική διαμαρτυρία γιατί είναι πάρα πολύ δυναμική σε ό,τι αφορά την πράσπιση των συμφερόντων τους. Αλλά το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι ότι οι μικροί γαλακτοπαραγωγοί βρίσκονται σε πολύ αδύναμη θέση στην αγορά. Η απάντηση της Γερμανίας ήταν ότι οι μικροί γαλακτοπαραγωγοί θα πρέπει να συμφωνήσουν να ε, συνδεθούν, αν θέλετε, σε μεγαλύτερους συνεταιρισμού. Αυτό έχει όμως και οικολογικές συνέπειες. Αυτό που είπε και ο συναδελφός Μπεζέτη σε κάποιον άλλο τομέα. Από οικολογικής άποψη, θα είχε νόημα να υπάρχουν μικρές εκμεταλλεύσεις και να διασφαλίσουμε τον καλύτερο, την καλύτερη ανταγωνιστικότητά τους προκειμένου να αποσυμπιεστεί κάπως η πίεση που στην οποία υπόκεινται. Και μάλιστα αυτό θα πρέπει να γίνει με τις τιμές της αγοράς, χωρίς επιδοτήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ήθελα να το θέσω ως διάσταση. Δεν είμαι κατά των άμεσων ενισχύσεων στην γεωργία, αλλά κάποιοι μικροί γαλακτοπαραγωγοί δηλώνουν ότι αυτό μεταφράζεται σε τιμές, μετακυλείται στις τιμές της αγοράς και ουσιαστικά δεν τους βοηθάει. Απλά διαμορφώνει με πολύ ύποπτο τρόπο τελικά τις τιμές στην αγορά. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό, Μάρκους. Έχει μία πτυχή που έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Θεωρώ ότι το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίσετε. Και εδώ πέρα κλείνω. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> προτιμάτε να κάνετε ιστορική συζήτηση, λέει ο κύριος Αλμούνια. Μάλιστα, κοιτάξτε. Να απαντήσω στο θέμα της Google. Είναι γνωστό ότι στα τέλη του 2010 ξεκίνησε μία έρευνα σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη παραβίαση του νόμου κατά τον τραστ στην αγορά της ηλεκτρονικής αναζήτησης στην Ευρώπη ιδιαίτερος. Ε, μονοπολεί ουσιαστικά η Google. Πάνω από το 90% του μεριδίου της αγοράς έχει η Google στον τομέα αυτό της αναζήτησης. Τέσσερα βασικά σημεία μας ανησύχησαν. Καταρχάς ο τρόπος με τον οποίο οι ανταγωνιστές της υπηρεσίας κάθε της αναζήτησης που προσφέρει η Google αντιμετωπίζονται και κατά πόσον υπάρχει σωστή εφαρμογή των ε, νόμων ε, για τον ανταγωνισμό, σε ό,τι αφορά δηλαδή την κάθετη αναζήτηση, αναζήτηση δηλαδή για εστιατόρια λοιπά, Για συγκεκριμένα ζητήματα. Και στην αγορά υπάρχουν ανταγωνιστές. Οι υπηρεσίες της Google Δεύτερη ανησυχία, ενδεχόμενη χρήση από την Google στα αποτελέσματα της αναζήτησης περιεχομένων άλλων, χωρίς ε, την συνένεση αυτών που έχουν παράγει το περιεχόμενο. Τρίτον, ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματεύτηκε η Google συμφωνίες με τις πλατφόρμες εκείνες με τους φορείς του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την μηχανή αναζήτησης ε, της Google συμπληρωματικά ως προ τις πληροφορίες που παράγουν και παρέχουν στο website τους. Και τέταρτον, οι όροι και με τους οποίους αντιμετωπίζει η Google το λογισμικό και αυτούς που παράγουν διαφημίσεις, ε, ανακοινώσεις στην πλατφόρμα του, της Google. Γιατί λάβαμε καταγγελίε καταγγελίες ότι το λογισμικό αυτό δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από άλλες πλατφόρμες από τους ίδιους ε, συντάκτες των διαφημίσεων αυτών. Ξεκινήσαμε λοιπόν τις σχετικές συζητήσεις και τώρα βρισκόμαστε στη φάση ανάλυσης των προτάσεων που μας υπέβαλε η Google πριν από κάποιους μήνες, προκειμένου να καθησυχάσει τις ανησυχίες μας, τις οποίες και επίσημα διαβιβάσαμε προς την Google. Βρισκόμαστε σε μια φάση δοκιμής της αγοράς. Υποβάλαμε την πρόταση της Google για να καθησυχαστούν οι ανησυχίες μας προς όλους τους φορείς και τους καταγγέλλοντες. Αυτή η δοκιμή για τις αγοράς ε, ουσιαστικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί χτες, αλλά κατόπιν αιτήματος κάποιων, των φορέ... κάποιων από αυτών των φορέων αποφασίσαμε να δώσουμε παράταση ενός μήνα. Τέλη Ιουνίου λοιπόν θα λάβουμε τις απαντήσεις αυτών που ενημερώθηκαν για τις προτάσεις της Google. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις απαντήσεις που λάβαμε. Θα ζητήσουμε από την Google κατά πάσα πιθανότητα, δεν μπορώ αυτό να το προεξοφλήσω ασφαλώς, αλλά είμαι σχετικά σίγουρος ότι θα, βοηθήσει, θα ζητήσουμε από την Google να βελτιώσει τις προτάσεις της. Και αν στα τέλη των ανταλλαγών αυτών η Google μας στείλει την πρόταση που θεωρούμε ότι καθησυχάζει τις ανησυχίες μας, θα εγκρίνουμε την απόφαση αυτή βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού, μεταφέροντας αν θέλετε, μεταφράζοντας αυτές τις προτάσεις σε νομικά δεσμευτικές δεσμεύσεις. Αν δεν τελεσφορήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να φτάσουμε τη διαδικασία του άρθρου 7 του κανονισμού μέχρι τέλους, με αρνητική απόφαση. Ελπίζω, ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια θετική λύση βάσει του άρθρου 9. Αυτό τι θα σημαίνει ότι μέχρι τα τέλη του έτους θα έχουμε επιλύσει τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τις ε, μηχανές αναζήτησης της Google. Έχουμε και, άλλα, και άλλες υποθέσεις σε ό,τι αφορά την Google. Όχι σε φάση επίσημης έρευνας, αλλά έχουμε λάβει επίσημη καταγγελία σε ό,τι αφορά κάποιες πτυχές του οικοσυστήματος Android. Το επεξεργαζόμαστε και αυτό το αίτημα. Έχουμε λάβει επίσημη καταγγελία, την εξετάζουμε. Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει αν θα ανοίξουμε ή όχι επίσημη έρευνα. Και έχουμε και κάποιες άλλες πτυχές που σχετίζονται με την Google όταν η Google εξαγόρασε την Motorola. Έχουμε κάποιες υποθέσεις άλλων εταιρείων που κατηγορούν την Motorola για κατάχρηση της θέσης της στην αγορά λόγω χρήσης συγκεκριμένων ε, συστημάτων τα οποία κατήχε η Motorola με τρόπο που θα ήταν αντίθετο προς ε, τους κανόνες και την νομοθεσία για το αντιτράστη. Για τους γαλακτοπαραγωγούς τώρα. 21ος αιώνα και μιλάμε και για ένα προϊόν το οποίο υπάρχει από τις απαρχές ε, του κόσμου μας. Η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε αυτόν τον τομέα, αλλά σύμφωνα με την συνθήκη θα πρέπει να εφαρμόζεται οι αρχέ αυτές λαμβάνοντα υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του κλάδου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον τομέα του γάλακτος, υποβάλαμε πρωτοβουλίε προσπαθώντας να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κλάδου και των αρχών που διέπουν την νομοθεσία για, την, τον ανταγωνισμό. Η εφαρμογή των κανόνων αυτών σε γενικές γραμμές είναι θέμα των εθνικών αρμόδιων αρχών, γιατί η αγορά του γάλακτος είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Δεν έχουμε ακόμα λάβει οποιαδήποτε τέτοια έτοιμα για να το κοιτάξουμε το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είχαμε ποτέ περιπτώσεις παραβίαση των νόμων για το τραστ. Σε γενικές γραμμές, η συζήτηση μεταξύ του αγροτικού κλάδου και της εφαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού είναι κάτι πολύ σημαντικό και όχι ιδιαίτερα απλό. Όπως είπατε, υπάρχουν αρχές που διαπούν την αγορά. Η μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ υποτίθεται ότι θα οδηγούσε στο δρόμο των μηχανισμών της αγοράς. Υπό τον όρο ότι οι μηχανισμοί της αγοράς αυτοί θα ε, ισχύουν, θα πρέπει να υπάρχει ο ανταγωνισμός, γιατί δεν υπάρχει αγορά χωρίς πολιτική ανταγωνισμού. Αν οι αρχές που διέπουν την αγορά εφαρμόζονται χωρίς πολιτική ανταγωνισμού, τι να σας πω, εγώ προτιμώ την παλιά ΚΑΠ. Και να σας ε, πω ότι ποτέ δεν υποστηρίζα την παλιά κοινή αγροτική πολιτική. Προτιμώ, την προτιμώ όμως. Την προτιμώ αυτή την πολύ καλά ορισμένη πολιτική από μια που δεν θα έχει κανένα κανόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η πρόεδρο. Όταν θα κάνει σημαντικέ ερωτήσεις θα πρέπει να λαμβάνει και σημαντικέ απαντήσει, Αλλά σα παρακαλώ, Γιώργεν, μιλήσατε παραπάνω από δύο λεπτά, όπω σα είπε ο Μάρκο. Μάρκο, τώρα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε κι εσεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω όμω τίποτα για τον τομέα τη ε, γαλακτοπαραγωγή. Χαίρομαι που θα έχουμε συνεργασία μεταξύ Βαβαρίας και Καταλωνίας την επόμενη περίοδο όπως ξέρετε από τον τομέα της, του ποδοσφαίρου, πέρα από την πλάκα όμως. Ε, συγγνώμη, αλλά σας ε, κερδίσαμε. Τέλεια. Να συγκεντρωθούμε λίγο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για θέματα για τις τράπεζες μας. Ε, είπατε πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση την εβδομάδα αυτή, αν σωστά έχω ενημερωθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια πρόταση για μια υπηρεσία η οποία θα ασχολείται με θέματα τέτοια τραπεζικής ε, εξυγίανσης και έχουμε και το 127.6 σε ό,τι αφορά την νομική βάση. Θέλω να μας πείτε πώς μια τέτοια υπηρεσία θα διαμορφωθεί πού θα εδρεύει για να παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα που προκύπτει. Ήμουν πάρα πολύ σύντομος, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και ανταγωνισμό, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις σχετικά με το ποδόσφαιρο. Εγώ προσπάθησα να ερευνήσω τι γίνεται με τον Χαβιέ Μαρτίνε για την Πάγια αλλά φοβήθηκαν πως υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Λοιπόν, για τις τράπεζες είναι αλήθεια ότι ανακοινώσαμε ότι θα στείλουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για να θέσουμε σε εκκίνηση έναν ενίο μηχανισμό εξυγίανσης τραπεζών για την Ευρωζώνη δεν αποτελεί έκπληξη για κανέναν, γιατί αυτό αποτελεί ένα από τα στοιχεία της Τραπεζικής Ένωσης, που εδώ και ένα χρόνο έχει λάβει την υποστήριξη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και πολλών άλλων και του Κοινοβουλίου. Μια Τραπεζική Ένωση. Δίχως έναν νέο μηχανισμό εξυγίανσης δεν λειτουργεί. Επομένως, χρειαζόμαστε αυτόν τον ενιαίο μηχανισμό. Από εκεί και πέρα, πώς θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός. Ακόμη δεν έχουμε εγκρίνει την πρότασή μας, επομένως δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες, ούτε εξαρτάται από μένα, δεν είμαι ε, σε ηγετική θέση για, τον, ε, κατάρτιση, για την κατάρτιση της πρότασης αυτής ε, και η γάμα δέλτα ανταγωνισμού είναι φυσικά σε συνεννόηση με τη γάμα δέλτα εκφήν και τη γάμα δέλτα για την ενή αγορά αν ε, ήμουν εγώ σε φντεφίλ θα μπορούσα να συζητήσω, αλλά δεν είμαι εμπειρογνώμονα στις νομικές βάσεις. Θα προσπαθήσουμε να λάβει πλήρη υποστήριξη από την ε, νομική μας υπηρεσία και ξέρω ότι σε διάφορα κράτη-μέλη γίνεται μία συζήτηση, από όσο γνωρίζω στη Γερμανία σίγουρα, σε σχέση με το εξής. Αν ε, απουσία μίας αναθεώρησης των συνθήκων, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια ενιαία αρχή εξυγίανσης ή αν ο μηχανισμός ε, θα πρέπει να είναι λιγότερο φιλόδοξος. Αλλά στη συζήτηση αυτή δεν θα μπω εδώ σήμερα. Θα το δούμε και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν ε, πριν να εγκρίνουμε την νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Επομένω, την επόμενη εβδομάδα δεν θα εγκρίνουμε την ε, πρωτοβουλία. Θα έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες εβδομάδες προς συζήτηση. Ευχαριστώ. Τα τελευταία χρόνια και το σχολιάσατε κι εσείς ε, όταν μιλήσατε για την αναδιάρθρωση και την εξυγίανση των τραπεζών. Το κάνατε αυτό ήδη σε προηγουμένα χαρτοφυλάκια. Γιατί λοιπόν χρειάζεται μια νέα υπηρεσία, ένας νέος οργανισμός. Εγώ ω Επιτρόπο Ανταγωνισμού είμαι υπευθυνό για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Όπω εξήγησα προηγουμένω στην κυρία Φερέιρα, μια διαδικασία τραπεζική εξηγίαση εν μέρη έχει να κάνει με τι κρατικέ ενισχύσει και το έχει να κάνει αυτό και με τον bailout, στην περίπτωση ενός bailout, ε, αμέσως χρησιμοποιούμε κρατικές ενισχύσεις, αλλά όταν μιλάμε για bail-in, διασημιδία μέσα δηλαδή, τότε εκεί δεν επισέρχονται οι κρατικές ενισχύσεις. Επομένως, αυτό που κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, είναι να δράσουμε ως μία αρχή εξυγένσης de facto, γιατί το μόνο μέσο εξυγένση που συνεισφέρει σε μια εξυγένση και διαθέτει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, το μόνο μέσο είναι το μέσο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων, αλλά δεν αρκεί. Και θα σας αναφέρω κάτι που γνωρίζετε εσείς πολύ καλά. Αν στην Επιτροπή ή οπουδήποτε αλλού στην Ευρωζώνη ε, ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε μία αρχή, απόφαση για την ε, αναδιάρθρωση της ΒΑΙΑΛΤ δεν θα είχε καθυστερήσει τέσσερα χρόνια. Τώρα το ΕΛΚ Πετικάινεν. Ευχαριστώ. Εδώ, εδώ. επεξεργαζόμαστε τη μεταρρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων τώρα στο Κοινοβούλιο και τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλω όμως να τονίσω, να σας ρωτήσω την άποψή σας για το ότι η Κομισιόν δαπάνησε πάρα πολύ χρόνο για ελάσσονα θέματα ενώ δεν έχει επαρκείς πόρους και τη δυνατότητα να αντιδράσει για τα κυριότερα θέματα για τις τρευλώσεις της αγοράς που μπορεί να προκαλούνται από ενισχύσεις όπως την αυπηγική και αλλού. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πρώτον τι ρυθμίσεις επεξεργάζεται η Κομισιόν ώστε τα ελάσσονα αυτά θέματα που <clears throat> αφορούν τη στήριξη μήκη όμικρων ή μικρών επιχειρήσεων να έχουν περισσότερους πόρους, να παρακαμφθούν και να δοθούν περισσότεροι πόροι στα κυριότερα θέματα. Thank you. Thank you Ευχαριστώ πολύ. είναι και αυτός ένας από τους στόχους που προσπαθούμε να επεξεργαστούμε στη στρατηγική εξυγχρονισμού σε τρία τουλάχιστον επίπεδα. Στην στον αναθεωρημένο διαδικαστικό κανονισμό Propose a simplified way. προτείνουμε έναν απλοποιημένο τρόπο για να χειριζόμαστε τα παράπονα και τις υποβολές και πολλές από αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε να λυθούν, να λύνονται πολύ σύντομα. Αλλά με την ισχύουσα διαδικασία δεν μπορούμε να επιταχύνουμε τις αποφάσεις γιατί εξαρτώμαστε από την απάντηση που θα δώσουν τα κράτη-μέλη κλπ. κλπ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η απλοποίηση της διεκπαιρέωσης αυτών των παραπώνων. Δεύτερον, μία γενική εξαίρεση όπου να διευρύνουμε τον τρόπο με τον οποίο να εφαρμόζουμε τις block exceptions και τι σημαίνει αυτός ο όρος ότι δεν θα ζητάμε εκ των προτέρων επαλήθευση ενός προγράμματος ώστε να επιτραπεί εθνικός να χορηγηθεί η στήριξη. Αυτή η ρύθμιση για τις block exemptions λοιπόν βρίσκεται στα πρώτα βήματα επεξεργασίας αλλά ελπίζουμε να εγκριθεί τέλος του 13 αρχές του 14 θα γνωμοδοτήσει φυσικά και το Κοινοβούλιο, θα το στείλουμε και στο Συμβούλιο και αν εγκριθεί όπως το προτείνουμε θα πάω και εγώ αύριο στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού όπου ελπίζουμε να εγκριθεί ο κανονισμός αυτός, η ρύθμιση αυτή τότε θα μπορέσουμε να διευρύνουμε το πεδίο της τομής όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ρύθμιση αυτή. στις ελάσσονες περιπτώσεις όπως είπατε και εσείς θα επιταχύνονται τα πράγματα για να ε, προσέξουμε περισσότερο τις ε, πιο σοβαρές περιπτώσεις. Αλλά για να γίνει αυτό το block exemption και να καταργηθεί εκ των προτέρων γνωστοποίηση χρειάζεται και ένα συνοδευτικό μέτρο δηλαδή η ενίσχυση εκ των υστέρων ελέγχου και το είχα πει και πριν από μερικούς μήνες εδώ στην μελέτη μας για το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια με τις αποφάσεις που είχαν ε, τύχει block exemption δεν είχαμε δηλαδή πρώτερη γνωστοποίηση βρήκαμε πάνω από ένα τρίτο των περιπτώσεων με λάθη στην δήλωση πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τις αρχές των κρατών μελών να είναι πολύ αυστηρές και ακριβής στον καθορισμό των προγραμμάτων και στην κατανομή των χρημάτων των φορολογουμένων γιατί δίνουν τα, τα κρατη δίνουν τα χρήματα και αν δεν εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις μας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε κι εμείς. Και τρίτον, μερικές αποφάσεις των κρατών μελών για επιχορηγήσεις δεν εγκρίνονται σε λογικό χρονικό διάστημα γιατί εξαρτόμαστε και εμείς από πληροφορίες που μόνο το κράτο μέλος μπορεί να μας δώσει. Και τα κίνητρα δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα γιατί σε μερικές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη προτιμούν να παρατείνουν την εξέταση του θέματος χωρίς να λαμβάνουν απόφαση ή δεν φροντίζουν επαρκώς να συλλέξουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε εμείς για να εγκρίνουμε μια απόφαση. Ζητούμε λοιπόν σε αυτή τη ρύθμιση να δοθεί η δυνατότητα υπό ορισμένες συνθήκες βέβαια να χρησιμοποιηθούν νέα εργαλεία αγοράς <laughs> μέσω εκείνων που κατέχουν τα στοιχεία αυτά άμεσα δηλαδή για να προετοιμάζουμε και εμείς σωστότερα το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ. Ε, τώρα ο Αντολίνη για το Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Εγώ λυπάμαι που για χρονικούς λόγους δεν μπορέσαμε να εγκρίνουμε τη δική μας έκθεση περί ανταγωνισμού μέχρι τη σημερινή συζήτηση. Θα ήθελα να πω ότι εμείς στην Επιτροπή Οικονομικών επαναλαμβάνουμε την πρόταση εξυγένσης ότι η αποζημίωση θα πρέπει να γίνεται μέσω ε, συλλογικών αλλά και ατομικών ε, Τώρα σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση είναι πολύ σημαντικό να διαρθρώσουμε καλά τη δράση της πολιτικής ανταγωνισμού με το θέμα της εξυγίανσης. Όταν χρησιμοποιούνται οι κρατικές ενισχύσεις πρέπει να υπάρχουν ίδιες πρώτερες συνθήκες για όλα τα κράτη-μέλη και να ισχύουν με τον ίδιο τρόπο για όλα τα κράτη-μέλη γιατί αλλιώ θα έχουμε κατακαιρματισμό. Και εγώ πιστεύω ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ε, θα πρέπει ε, να παρουσιαστούν όταν υπάρχει και ο κανονισμός εξυγίανσης και σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις. Τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε 1.400 αποφάσεις περί κρατικών ενισχύσεων και από το 1 δέκατο οδήγησαν ε, σε διαδικασίες έρευνας ε, και το πέμπτο τμήμα σε επιστροφές. Έτσι λοιπόν ε, το πόσο κράτησαν ε, οι έρευνες και οι φάκελοι πολλές φορές ήταν ε, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παραδείγματο χάρη για την περίπτωση της Ισπανίας έχουμε μια έρευνα που διαρκεί δύο χρόνια και αυτό είχε συνέπειες ήδη πάρα πολύ αρνητικές για την περίπτωση των εναυπηγείων. Έτσι, λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε ποιο τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ, Αντολή. Όπως γνωρίζετε, εγώ προσωπικά και η Επιτροπή ήμασταν ε, υπέρ ε, του να ρυθμίσουμε όχι μόνο ε, την ατομική αλλά και τη συλλογική αποζημίωση. Ήταν ε, συλλογική απόφαση του Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια και είπε στην Κομισιόν ε, να μας στέλνετε ένα ε, νομοσχέδιο ενώνοντας και τα δύο. Εγώ δυστυχώς στεναχωρήθηκα, δεν μου άρεσε καθόλου. Το σέβομαι. Σέβομαι φυσικά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά δεν μου άρεσε η απόφαση του Κοινοβουλίου. Αλλά δεν ήταν δική μας απόφαση αυτή. Ήταν απόφαση που ήρθε από το Κοινοβούλιο, Τραπεζική Ένωση. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας στο ότι οι μηχανισμοί εξυγίανσης και για την Ευρωζώνη και για τις χώρες που συμμετέχουν αλλά και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν θα πρέπει να είναι τόσο ευέλικτος ώστε να δημιουργήσει προς τις τρευλώσεις στην εσωτερική αγορά και η κρίση έχει δημιουργήσει αρκετές στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά ε, από τα ασφάλιστρα κινδύνου μέχρι το κατακαιρματισμό του διατραπεζικού τομέα ή τις μεταβιβάσεις ρευστότητα μεταξύ οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο τραπεζικό όμιλο. Και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Και ο μηχανισμός εξυγίανσης τόσο για τους 27-28 όπως και για τους 17 συν δεν ε, θα έπρεπε να συμβαλεί σε αυτό και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα βοηθήσει την Κομισιόν να καταπολεμήσει αυτό τον κατακαιρματισμό γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες ε, που λαμβάνω για τη συνομοθετική διαδικασία δεν είναι και τόσο θετικά τα πράγματα. Μου δίνει την εντύπωση ότι στο Συμβούλιο οι βαθμοί της ευελιξίας καθημερινά αυξάνονται για τις ε, κρατικέ ενισχύσει, αποκλειστική αρμοδιότητα τη Κομισιόν. Θα πρέπει να διατηρηθούν κρατικέ ενισχύσει, θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι κανόνε για όλους και θα το κάνουμε στο βαθμό που νομίμω είναι δυνατό και στο βαθμό που δεν υπάρχει καινούργια νομοθεσία πρέπει να κάνουμε αυτά που ισχύουν. Αν εσείς ψηφίσετε μια νέα νομοθεσία με το Συμβούλιο και μας βοηθήσετε στο να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία θα προσπαθήσουμε ε, και πάλι να δράσουμε αλλά σεβόμενη μια βασική αρχή, την αρχή της μη διάκρισης. Τώρα η διάρκεια των φακέλων. Δεν ε, μπορώ να σας πω αυτό, δεν είναι ευθύνη της Κομισιόν. Εσείς ε, μαζί με το Συμβούλιο είστε δημοσιονομική αρχή, δεν μας δίνετε περισσότερους πόρους, μας δίνετε λιγότερους. Και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί έχουμε τεράστιο φόρτο εργασίας ε, που θα μπορούσε να απασχολήσει ένα χ της 100 παραπάνω στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και αυτό με πάρα πολλές ώρες δουλειά για τα καρτέλ, για τις συγχωνεύσεις, για τα διδράσεις, τις κριτικές ενισχύσεις κτλ. Δηλαδή αυξάνεται συνεχώ η συζήτηση και ο αριθμός των αποφάσεων που αναφέρεται ενελύεται από το 1 τρίτο τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ενώ τα άλλα δύο τρίτα εργάζονται σε άλλου τομεί και εκεί είναι πολύ μεγάλο το άχθο εργασία. Όμω δεν πρόκειται μόνο για περιορισμό των ανθρώπινων πόρων και την ικανότητα εργασία τη ΓΔΑ ανταγωνισμού στην περίπτωση κριτικών ενισχύσεων. Αν το κράτο μέλο δεν συνεργάζεται, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και εσείς ε, μου αναφέρατε το παράδειγμα του Ισπανικού προγράμματος που τέθηκε σε λειτουργία στην Ισπανία στις αρχές του 2002 και δεν κοινοποιήθηκε. Αν ε, είχε κοινοποιηθεί εκείνο το σύστημα εδώ και 10 χρόνια, θα το είχαμε λύσει αυτά τα πράγματα εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί. Τώρα, επειδή έφτασαν σε εμά μία σειρά παραπώνων που πρέπει να τα αναλύσουμε και να απαντήσουμε, μία σειρά καταγγελιών, ανοίξαμε την έρευνα εδώ και λιγότερο από δύο χρόνια και είμαστε πολύ κοντά στην τελική απόφαση. Σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους θα αρέσει λιγότερο. Όμω είμαστε κοντά στη λήψη τη τελική απόφαση, αφού καταβάλαμε πάρα πολλέ προσπάθειε εμεί ω Κομισιόν, για να μπορέσουμε να έχουμε στη διάθεσή μας απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη της απόφασης. Εγώ όταν διαβάζω τον ισπανικό τύπο, λέει ότι ο Αλμούνια καθυστερεί την απόφαση και λέω αυτός που πρέπει να υπογράψει, ναι είναι ο Αλμούνια, αλλά δεν ευθύνομαι εγώ για τους λόγους της καθυστέρησης, σας διαβεβαιώ. Καλά. Λάγκεν. Σας ευχαριστώ Επιτροπέ. Θα ήθελα να σας επενέσω για το συνολικό σας έργο. Κατά το παρελθόν ε, ε, τηρήσατε σε υψηλά επίπεδα την πολιτική για τον ανταγωνισμό παρά την, ε, τις εθνικές διαμαρτυρίες. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πω προκαταρτικά. Ήθελα να σας πω το εξή. Καταρχάς μιλήσατε για τις ε, καταθυντήριες γραμμές, για τα πολλά εθνικά αεροδρόμια τα οποία, τις οποίες θα παρουσιάσετε συντόμως. Πώς, ε, σε τι φάση βρίσκονται αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές πότε θα ολοκληρωθούν. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση, ευρυζωνική διασύνδεση των, ε, της υπαίθρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποίησε δημόσια κονδύλια. Πώς ε, προχωράει αυτή η υπόθεση όμως, σε τι φάση βρισκόμαστε. Και τελευταία ερώτηση σε ό,τι αφορά το Lobo Green, το οποίο το γνωρίζετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσε να αποδεχτεί αυτές τις κρατικές ε, ενισχύσεις. Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στην εξής φάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιτρέπει να παραμείνει η κατάσταση και οι υπόλοιπες ε, ε, επενδύσεις πάνω από 340 δισεκατομμύρια ευρώ να επιτραπούν. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν επιμένει να υπάρχει μια κλειστή διαδικασία. Εγώ με τις εμπειρίες που έχω στην πολιτική ανταγωνισμού δεν μπορώ να φανταστώ ότι ε, ισχύει όντω αυτό που αναφέρετε. Θεωρώ ότι είναι η δικαιολογία αυτή που προβάλλεται. Πείτε μου αν θέλετε και αν δεν μπορείτε να απαντήσετε σήμερα, ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε μια γραπτή απάντηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό στην ε, αντιπαράθεση. Ευχαριστώ κύριε Λαγκέλ, ευχαριστώ για τα αρχικά σας σχόλια. Να απαντήσω στις τρεις σας ερωτήσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές, για τις αεροπορικές εταιρείε και τα αεροδρόμια. Βρισκόμαστε σε διαδικασία διαβούλευσης, ελπίζω να μπορέσουν να εγκριθούν πριν τα τέλη του έτους. Τώρα, όταν θα εγκριθούν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την επίλυση το συντομότερο δυνατόν στις περίπου 60 υποθέσεις που κρεμούν για θέματα κρατικών ενισχύσεων, είτε πρόκειται για αεροδρόμια, είτε για εταιρείε αερομεταφορών που έχουν λάβει ενίσχυση επειδή πετούν σε ορισμένα αεροδρόμια. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνεχώ αναβαλόταν για δύο λόγου. Τρει. Γιατί υπάρχουν πολλά δημόσια κονδύλια και στις επενδύσεις και στην λειτουργία των περιφερειακών αεροδρομίων όπως ε, και στο να πετούν κάποιες εταιρείες σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Δεύτερον, καθυστέρησε γιατί υπήρξε από την ε, γάμα δέλτα μεταφορών, μία μεταφορά αρμοδιοτήτων. Στην γάμα δέλτα ανταγωνισμού έφτασαν πάρα πολλοί φάκελοι, αλλά ε, δεν είχαμε προσωπικό, δεν ήρθε κανένας και όλοι έπρεπε να μάθουν από την αρχή. Έτσι λοιπόν, ε, τώρα... Έχουμε φτάσει σε θέση να εγκρίνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές και να επιλύσουμε τις υποθέσεις. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι οι ισχύουσες κατευθυντηρίες γραμμές δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Αν τις εφαρμόζαμε, έτσι όπως είχαν εγκριθεί πριν πολλά χρόνια, θα έπρεπε να θετήσουμε αρνητικέ περιπτώσεις με ανάκτηση σε πολλές από αυτές τις 60 υποθέσεις και νομίζω ότι δεν είναι λογικό να το πράξουμε. Γιατί η χρήση ε, εταιριών χαμηλού κόστους ε, και σε περιφερειακά αεροδρόμια σε πολλές περιπτώσεις ότι ελογείται πλήρως. Επομένως υπάρχει ένας λόγος ουσιαστικός, όχι μόνο ανθρωπινών πόρων ή χρήση δημοσίου χρήματο. Δεύτερον, για τα ευρυζωνικέ υπηρεσίες. Εγκρίναμε τις νέες κατευθυντήριε γραμμές πέρσι το Δεκέμβριο και στο νέο κανονισμό διευκόλυνση έχουμε τη δυνατότητα εξαίρεση σε κατηγορία. Αν αύριο το Συμβούλιο δώσει το πράσινο φω και να υποστηρίξει και το Κοινοβούλιο, έχουμε ακόμη χρόνο να συμπεριλάβουμε το νέο κανονισμό αυτή την ε, προσθήκη που θα εγκριθεί από το Συμβούλιο στο νέο κανονισμό. Και τρίτο, για αυτό το ring που αναφερθήκατε. Μιλήσαμε και γραπτός ε, και προφορικά. Εγώ υπέγραψα χτες δύο επιστολές απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων και αμφιβαλιών που προήλθαν ε, από την ε, αρμόδια αρχή του Λάντ της Ρενανίας αλλά και από τον επενδυτική και εγώ απάντησα στις ερωτήσεις και στις ενσυχίες σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει για να εφαρμοστεί η απόφαση που θετήσαμε πέρσι. Γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, λέει η Πρόεδρος. Ναι, μία ερώτηση. Μιλάμε για guidelines ή για οδηγία σε ό,τι αφορά τα αεροδρόμια και κατά δεύτερον, αυτά τα έγγραφα είναι προσβάσιμα. Αν ε, εσείς μου στείλετε μια γραπτή ερώτηση, σας απαντήσω αυτά που μπορώ να σας απαντήσω. Ή αν έχουμε μια συνομιλία, ό,τι προτιμάτε. Αλλά δεν είναι δημόσια επιστολή. Μιλάμε για κατευθυντήριες γραμμές για τα αεροδρόμια και τις εταιρείε αερομεταφορών. Guidelines. Μακάρθη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Επίτροπε, να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για το έργο που κάνετε σε ό,τι αφορά labor και σε ό,τι αφορά τις έρευνες και τις ε, τιμές του πετρελαίου. Θα θυμάστε ότι σας έγραψα μετά από το ΙΟΣΚΟ που ε, έκανα έκθεση για ενδεχόμενη παραποίηση και σε ό,τι αφορά τις τιμές ε, των, ε, του αερίου. Γιατί ήρθε και μου κατέγγυλαν στο γραφείο μου ότι ε, έχασε κάποιο τη δουλειά του όταν βγήκε και μίλησε για τα στοιχεία αυτά, γιατί μιλάμε για 3 εκατομμύρια σε ό,τι αφορά και τα παράγωγα που εμπλέκονται. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξή: Αν αποδεχτεί ότι υπήρξε όντω παραποίηση και φυσικά υπάρχει αυτό το μεγάλο αν το οποίο θα προκύψει από τις έρευνες, θα υπάρξουν ε, πρόστιμα κυρώσεις. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Αλλά αυτό που με ανησυχεί και ορίζω την ιδέα του, της νομοθεσίας για την ιδιωτική εφαρμογή. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα έχει αναδρομική ισχύ αυτό. Και έχετε δίκιο. Και εγώ είχα ζητήσει αποζημιώσεις μετά την Virgin και την ε, British Airways που ε, είχαν ορίσει τιμές για τις διατραντικές πτήσεις και σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Συλλογική αγωγή έγινε στη Μεγάλη Βρετανία γιατί το επιτρέπει ο νόμος και με ανησυχεί λοιπόν το γεγονός ότι ό,τι και να γίνει στον τομέα αυτό δεν θα αποζημιώσει τον ε, καταναλωτή. Γιατί δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ η νομοθεσία. Θα μπορούσατε λοιπόν να γράψετε προς τα εθνικά κρατημέλη που είναι υπό έρευνα και να τα παροτρύνετε να εξετάσουν ενδεχόμενους τρόπους αποζημίωσης μέσω του εθνικού δικαίου του καταναλωτή. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα ένδικα μέσα. Νομίζω ότι όταν ολοκληρώσετε τις έρευνες αυτές θα έχετε στα χέρια σας πολύ λεπτομερή, ε, πολύ λεπτομερή στοιχεία για τις ε, πρακτικές για τα συστήματα που οδήγησαν στην παραποίηση των βασικών αυτών στοιχείων. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω ότι πέρα από την ε, νομοθεσία για το benchmark που είναι στον τομέα του Επιτρόπου Μπαρνιέ θα συνεχίσετε τις διαβουλεύσεις για να διασφαλίσετε και να δούμε πώς μπορούμε στο μέλλον να αποφύγουμε αυτό που είναι δική σας ευθύνη. Να αποφύγουμε τέτοιες δομές που δεν είναι ανταγωνιστικές, που έχουν σύγκρουση συμφερόντων. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ η απάντηση. Δεν πιστεύω ότι κάποια νέα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την διαδοκή εφαρμογή των ε, παραβιάσεων του νόμου περί ανταγωνισμού μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ. Δεν νομίζω ότι τέτοια νομοθεσία μπορεί ποτέ να έχει αναδρομική ισχύ, αλλά όπως είπατε σε κάποια από τα κρατημέλη υπάρχει τέτοια νομοθεσία και μάλιστα υπήρχε και πριν τα περιστατικά αυτά ή μάλιστα ίσως παράλληλα με, την, ε, με τα περιστατικά αυτά και φυσικά σε εθνικό επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μέσα αυτά. Αυτό δεν είναι όμως δικό μου καθήκον. Δεν μπορώ να πω εγώ στα κρατημέλη πώς θα χρησιμοποιήσουν τις αρμοδιότητες τους. Θα μπορούσατε όμως να, να αποκαλύψετε τα αποτελέσματα των ερευνών σας. Ναι, κοιτάξτε, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν γιατί οι έρευνες προχωρούν και όλα αυτά τα πορίσματα των ερευνών θα είναι δημόσια. Αλλά βρισκόμαστε στην αρχή της έρευνας. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλος, δεν έχουμε φτάσει στα πορίσματα. Σε ό,τι αφορά τα ενδικά μέσα, όπως είπατε, ο Μισελ Μπαρνιέ ως επίτροπο για την Ιστορική Αγορά είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να προτείνει μια νέα τέτοια νομοθεσία για τον ορισμό των benchmarks αυτός, αυτών. Και άλλες ε, δικαιοδοσίες εμπλέκονται σε εθνικό επίπεδο, είχα επαφή με τις Βρετανικές Αρχές ε, και σε επίπεδο κοινοβουλίου έγιναν ε, σεμινάρια που τριγανώθηκαν από το κοινοβουλίο δηλαδή. δηλαδή και από τη γενική μου διεύθυνση συμμετέχουμε απόλυτα στο νομοθετικό αυτό έργο και συμβάλλουμε ωστόσο σε περιορισμένο βαθμό γιατί γνωρίζουμε σε όλη την έρευνα ότι όλα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά απόρριτα. Αλλά όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν χρειάζεται να παραμείνουν απόρριτα ασφαλώς και θα τα χορηγήσουμε. Ελπίζω έτσι να συμβάλλουμε με επικοδομητικό τρόπο για να πετύχουμε μια καλή νομοθεσία που χρειάζεται σε όλα τα benchmarks. Ξεκινήσαμε στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Τώρα είμαστε στον κλάδο της ενέργειας και κατά πάσα πιθανότητα και σε διαφορά τον κλάδο των πρώτων υλών θα πρέπει να προσέξουμε. Ναι, ναι, ναι, όχι όμως τόσο, δεν είμαστε τόσο προηγουμένοι σε τόσο προηγουμένη φάση όπως στον τομέα του πετρελαίου. Μάλιστα λέει η Πρόεδρος, σίγουρα και το θέμα των πρώτων ε, υλών θα τεθεί. Ο Πάμπλο από το ΕΛΚΑ. Panic. I will use this one. Uh, uh, Ευχαριστώ, Επίτροπε. Αν ε, θέλατε να ερευνήσετε την περίπτωση της χώρας μου, Μαρτίνετε, θα θέλατε, ελπίζω, να <laughs> ερευνήσετε και την περίπτωση της Ατλέτικο. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ξεχωριστή υπόθεση. Τώρα όμως, ε, για να μπούμε στα νομοθετικά. Τρεις σύντομες ερωτήσεις ε, για το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόστηκε για την κατασκευή ναυπηγείων ε, στην Ισπανία. Υπήρχαν διάφορα εκεί, διάφορες συνιστώσεις επιλεξιμότητας. Ε, η Ισπανία χρησιμοποίησε ένα νέο καθεστώς που εξαλείφει κάθε συνιστώς επιλεκτικότητας. Όμως, παρόλα αυτά, υπάρχουν άλλες χώρες όπως η Ολλανδία που χρησιμοποιεί διάφορες συνιστώσει, επιλεξιμότητε και έγινε σχετική καταγγελία στην ΓΔ ανταγωνισμού και συνεχίζω, ο μιλητής χωρίς μικρόφωνο. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε αν έχουν ανοίξει έρευνες για αυτά τα θέματα. Δεύτερον, για το πειθαρχικό καθεστώς της Κομισιόν για τα καρτέλ. Αυτό συμπεριλαμβάνεται σε ένα μη νομοθετικό εργαλείο στις κατευθύνες γραμμές του 2006. Πιστεύετε ότι δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη βεβαιότητα σε όλη τη διαδικασία, αν είχαμε ένα κανονισμό αντί για αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές, όπως είπε και το Κοινοβούλιο σχετικά με την εκ της ανταγωνισμού. Και τρίτον, η εφαρμογή κυρώσεων για πρακτικές ε, καρτέλες επιχειρήσεις που παράγουν ένα προϊόν και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προσφέρει προβλήματα λόγω των ε, ιδιότυπων στοιχείων. Δεν πιστεύετε ότι αυτό το σύστημα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ε, που παράγουν ένα και μόνο προϊόν να το εισβάλλεται στις κατευθυντήριες γραμμές αντί να γίνεται αξιολόγηση αναπερίπτωση. Επίτροπος, ευχαριστώ να σας πω κάτι που δεν θα έπρεπε να μπει στα πρακτικά της συνεδρίασης, αλλά οποιαδήποτε οικονομική σχέση ε, σε σχέση με αυτό το θέμα ανήκει στην αρμόδια αρχή ανταγωνισμού της Ισπανίας. Τώρα για το ταξιλής. Υπάρχουν συστήματα ταξιλής ε, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες στις ε, κατευθυντήριες γραμμές για τον τομέα της ναυτιλίας Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν δηλωθεί συμβατά για αυτό το τομέα. Παραδείγματο ε, χάρη ο φόρο χωρητικότητας ή τα ειδικά χαρακτηριστικά για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ε, για τους εργαζομένους, ε, για τα πληρώματα στα σκάφη. Υπάρχουν λοιπόν πολλά συστήματα τέτοιου είδους που μπορεί να είναι συμβατά. Υιοθετήσαμε μάλιστα και μία απόφαση δηλώνοντας συμβατό το νέο ισπανικό σύστημα. και δεν αναφέρεται μόνο στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά χρησιμοποιήθηκε βασικά για τον ναυτιλιακό τομέα. Δεν είναι όμως επιλεκτικό. Είδαμε και άλλες συστήματα και άλλες χώρες, ναι, ξεκινήσαμε έρευνες επίσημα για άλλα συστήματα άλλων κρατών μελών πέρα από την ισπανική περίπτωση και όπως είπατε λάβαμε μια καταγγελία από την Ισπανία για το Ολλανδικό σύστημα και το εξετάζουμε. Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν θα υπάρξει έναρξη ή μη ερευνητικών διαδικασιών, αλλά φυσικά εργαζόμαστε επί αυτού του ζητήματος. Δεύτερον, για τα πρόστιμα στην περίπτωση καρτέλη ή αντιτράστ. Εγώ ξέρω ότι το Κοινοβούλιο ενίοτε έχει ζητήσει από την Κομισιόν να συμπεριλάβει τις προβλέψεις και τα κριτήρια που έχουμε στις κατευθυντήριες γραμμές για τα πρόστιμα του 2006 σε ένα κανονισμό. Εμεί πιστεύουμε ότι δεν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Κατανοώ το Κοινοβούλιο να ζητά να νομοθετήσουμε, είναι λογικό. Όμως και εγώ νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της ε, διαδικαστικής οικονομίας και αν μπορούμε να λύσουμε κάποια στιγμή χωρίς να προσφύγουμε ε, σε νομοθετική διαδικασία που ξέρετε είναι πολύ πιο βαριά γιατί στη συνέχεια είναι πολύ πιο δύσκολη η τροποποίηση μπορούμε να προσφεύγουμε πολύ καλά στις κατευθυντήριες γραμμές. Ήδη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου έχει λάβει κάποιες αποφάσεις που υποστηρίζουν τις σημερινές κατευθυντήριες γραμμές και μας δικαιώνει στις περιπτώσεις που έχουν εφαρμοστεί. Για το τελευταίο θέμα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που παράγουν ένα μόνο προϊόν, χωρίς να υπάρχει αναγκαιότητα να αναφέρεται αυτό ρητός στις κατευθυντήριες γραμμές, υπάρχει τουλάχιστον μια απόφαση για τα καρτέλ που λαμβάνεται υπόψη τη στιγμή που καθορίζεται το ύψος ε, των ε, προστήμων, ε, το αν υπάρχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που παράγουν ένα και μόνο προϊόν. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Αναπτυμεσία. Η Μαρλίν είναι η νέα αντιπρόεδρος που αντικαθιστά τον Έντουαρτ Σικλούνε, ο οποίος ε, διορίστηκε υπουργός οικονομικός στη Μάλτα, όπως γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ. Επίτροπε, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους ε, ζητήσατε να καταρτιστεί η νομοθεσία σε ό,τι αφορά περιπτώσεις κακοδιαχείρισης. Αυτό έγινε αποδεκτό με μεγάλη πλειοψηφία και καταλαβαίνετε φυσικά πόσο σημαντικό είναι αυτό για το θέμα του ανταγωνισμού. Σας ερωτώ λοιπόν το εξή σύντομο ερώτημα. Γιατί δεν έχει κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση δηλαδή ε, της, των δομών της αναδιάρθρωσης των εταιριών. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι στον τομέα των αρμοδιοτήτων μου. Ίσως είναι θέμα εσωτερική αγοράς. Εκπροσωπείτε το κολέγιο των επιτρόπων, το σώμα των επιτρόπων εδώ. Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν έχω απαντήσει σε όλα τα πιθανά ερωτήματα με όλο το σεβασμό που σα τρέφω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα και στο ερώτημα αυτό μπορώ να το ε, διαβιβάσω στον Μισελ Βαρνί, τον συνάδελφό μου που είναι ο αρμόδιο νομίζω για τέτοια θέματα. Το ίδιο και Είπα και στον κύριο Κοζές, δεν μπορώ να απαντήσω επί παντός επίστητου. Είναι χιλιάδες θέματα. Κοιτάξτε όμως, δεδομένη στη σημασία στις νομοθεσίας και του τρόπου που ψηφίστηκε, κοιτάξτε, θα πρέπει να διαβιβάσω στο Μισελ Μπαρνιέ το έντονο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν υπάρχουν πολλά θέματα που δεν μπορεί να τα αναφέρει δημόσια φαίνεται. Λοιπόν, Τελευταίο ερώτημα από τους φιλελεύθερους Σμιτ. Περίμενε υπομονητικά. Σας κατευχαριστώ. Ξέρω ότι είστε σοφός άνθρωπος κύριε Επίτροπε, άρα εμένα θα μου απαντήσετε λοιπόν για τις τιμές της ενέργειας. Τα συμπεράσματα του προηγούμενου Συμβουλίου προέβλεπαν πολλές ad hoc δραστηριότητες. Άκουσα χθες ότι η BMW κατασκευάζει ένα καινούργιο εργοστάσιο εκτός Γερμανίας γιατί είναι πολύ ψηλές οι ενεργειακές τιμές εκεί και υπάρχει και η επανάσταση εδώ τώρα των, του σχιστολιθικού αερίου κλπ. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι καιρό είναι να υπάρξει ένα κοινό σχέδιο δράσης για τα ενεργειακά γιατί εδώ χάνουμε ανταγωνιστικότητα. Αυτό ήταν η πρώτη ερώτηση. Υπάρχει όμως και δεύτερη. Άκουσα επίσης φήμες ότι μέσα στην Κομισιόν συζητάτε μέτρα και για τη χαλιβουργία λέει. Μπορείτε να μου διασφαλίσετε για να μην μπομάσει γιατί είμαστε πολύ λίγοι ότι αυτά τα μέτρα και τα σχέδια για τη χαλιβουργία στην Ευρώπη θα ευθυγραμμίζονται με την πολιτική ανταγωνισμού της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σμίτ. Για την ενέργεια διάβασα και εγώ με πολύ ενδιαφέρον και πολύ προσοχή τα συμπεράσματα του προηγούμενου Συμβουλίου για, την, για τα ενεργειακά γιατί είχα πει και στην αρχική μου παρουσίαση ότι από την άποψη του ανταγωνισμού και ως προς την καταπολέμηση των τραστ και καρτέλ και ως προς τις κρατικές επιχορηγήσεις φάνηκε ότι κάθε μέρα τίθενται ενεργειακά προβλήματα. Είναι ένας τομέας πάρα πολύ σημαντικός για όλη μας την οικονομία και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι κανόνες του ανταγωνισμού να εφαρμόζονται σωστά. Για την επανάσταση του σχιστολιθικού αυτή μας θέτει ένα μεγάλο, μια μεγάλη πρόκληση. Όταν διάβασα τα συμπεράσματα αυτά χάρηκα ιδιαίτερα γιατί οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είπαν επιβεβαιώνουμε τη θέλησή μας να προχωρήσουμε προς ενιαία εσωτερική αγορά ενεργείας για του χρόνου. Ταυτόχρονα όμως, επειδή συνήθως έτσι λένε τα συμπεράσματα, Θέλησα να δω και πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερες διασυνδέσεις και δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να υπάρχει ενιαία αγορά ενεργείας στην Ευρώπη χωρίς πραγματική σύνδεση των αγορών σε ολόκληρη την Ευρώπη και στο αέριο και στον ηλεκτρισμό. Αν δω λοιπόν τι άλλο κάνει η Ένωση ας πούμε το επόμενο Πολδίπ και το Connecting Europe. Πώς θα συνδέονται όλα αυτά με την ενέργεια. Εκεί βρήκα ότι δεν υπάρχει τίποτα σχεδόν. Πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν τρόπο να χρηματοδοτήσουμε τεράστιες επενδύσεις και να βρούμε τρόπο επίσης να αποφασίσουμε πολιτικά πώς θα καταλήξουμε σε πραγματικές διασυνδέσεις μεταξύ ας πούμε αερίου και ηλεκτρισμού. Προηγουμένως με ρώτησε ο κύριος Λεσέντ για τη στήριξη των ανανεωσίμων. Αν δεν το συνδέσουμε και αυτό με τα υπόλοιπα, κάποια μέρα θα χρειαστεί να μειώσουμε τη στήριξη των ανανεωσίμων. Γιατί η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να ούτε να αποθηκευτεί ούτε να σταματήσει και αυτό θα κατέληγε λοιπόν σε σπατάλη δηλαδή ενεργειακός πόρος που δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χώρα όπου παράγεται ούτε να μετασχηματιστεί σε άλλη μορφή. Τέλος. Το energy mix με ή χωρίς πυρηνικά, με ή χωρίς περισσότερα ανανεώσιμα, με ορυκτά καύσιμα έχουμε πολλή δουλειά για να συνδέσουμε όλα αυτά με τις κρατικές βοήθειες ή με τα μέτρα αντιτράστ. Όλα αυτά πρέπει να τα συνδυάσουμε. Αλλιώς, από τη μία τα σκιστολιθικά, από την άλλη το φυσικό, από την άλλη οι αναδιόμενες με την ανταγωνιστικότητά τους. Αφού μιλάμε για ανταγωνιστικότητα και για 20% περισσότερη εκβιομηχάνηση το 20 και σε 20 χρόνια δεν θα είμαστε πια ανταγωνιστικοί με καμία περιοχή του κόσμου αν δεν σοβαρευτούμε σε αυτόν τον τομέα την ενέργεια. Εγώ ως Επίτροπος Ανταγωνισμού κάθε μέρα μελετάω τις επιπτώσεις που έχει η έλλειψη της κοινή στρατηγικής για όλα αυτά. Για την Χαλιφούργια, από ό,τι γνωρίζω, για τις προτάσεις του συναδέλφου μου Ταγιάννη, σε συνεννόηση βέβαια με τους ενδιαφερόμενους τομέα κλπ. Σε κανένα από τα τμήματα της στρατηγικής για το Χάλιβα δεν βλέπουμε λόγο να διστάσουμε. Αλλά ας μην συνεχίσω γιατί ξέρετε. Ο Λάγκεν νικετεύει να λάβει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, να σας παρακαλέσω αν είναι δυνατόν να απαντήσετε και στη τρίτη ερώτηση που σας έθεσα σε ό,τι αφορά την ευρυζωνική διασύνδεση στην Ήπετρο και σε ό,τι αφορά και ό,τι αφορά τις δημόσιες ε, επιδοτήσεις. Υπάρχουν απαλλαγές, εξαιρεσει. Ε, ε, δεν ξέρω κατά πόσον μήπως επεξεργάζεται τους σχετικούς κανόνες. Αν έχετε την ευκαιρία και το χρόνο να μου πείτε προς το... Να μου πείτε πόσο έχετε επεξεργαστεί αυτά τα θέματα σε ό,τι αφορά τους τομεί τη βιομηχανία που είναι υψηλή σε κατανάλωση ενέργειας. Okay. Νομίζω ότι απάντησα στην προηγούμενη παρέμβαση μου για τα ευρυζωνικά. Τέλος πάντων, θα επαναλάβω. Υιοθετήσαμε τις νέες κατευθυντηρίες γραμμές για τα ευρυζωνικά πέρσι το Δεκέμβριο. Τώρα, εξετάζουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Αν στον ε, νέο κανονισμό που θα συζητηθεί αύριο σε επίπεδο Συμβουλίου. Υποστηριχτεί δική μου θέση να διευρυνθεί να διευρυνθούν οι, δυνατότητες ε, των επενδύσεων block exempting, τότε αυτό μπορεί να μπει στο γενικό κανονισμό block exceptions που θα πρέπει να υιοθετηθεί στα τέλη του έτους ή αρχές του 2014 αλλά και στο δικό μας κανονισμό της Κομισιόν χρειάζομαι την έγκριση από τον κανονισμό του Συμβουλίου. Τώρα, για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ιδίως για τη Γερμανία, αλλά όχι μόνο. Έχουμε ένα σύστημα που είχε προετοιμαστεί στη Γερμανία το 2009, για να αποζημιωθούν κάποιοι τομείς ε, για την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα μπορεί να αυξήσουν το κόστος αυτών των εργοβόρων βιομηχανιών. Σταματήσαμε την έρευνα για αυτό το θέμα, γιατί προετοιμάζαμε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές ε, για το ETS, ε, το σύστημα εκπορίας εκπομπών, αλλά νομίζω ότι η συμφωνία στην οποία θα καταληξούμε θα είναι πολύ καλή και ήταν πολύ καλή και ισορροπημένη, γιατί όλοι ήταν ικανοποιημένοι με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές ETS. Έχουμε ξεκινήσει μία έρευνα στη Γερμανία για τη μεταχείριση από τη σκοπιά του χειριστή ε, του δικτύου γιατί υπάρχει μια εξαίρεση για ορισμένες τέτοιες ενεργοφόρες βιομηχανίας ε, που χρηματοδοτούνται από τους άλλους χρήστες του διαχειριστή δικτύου και υπάρχουν επιβαρύνσεις που μεταβάζονται στους καταναλωτές. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την έρευνα και το αναλύουμε το θέμα, εξετάζουμε το αν θα ξεκινήσουμε μια έρευνα ή όχι, αν θα ανοίξουμε έρευνα για το άλλο γερμανικό σύστημα που ισχύει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πάνω κάτω υπάρχει διαμεταχείριση. Με την περίπτωση των ενεργοβαρομηχανιών δεν έχουν καταβάλει ε, τις ε, επιπλέον χρεώσεις ή πληρώνουν πάρα πολύ χαμηλά τέλη και τελικά είναι οι καταναλωτές αυτοί που πληρώνουν το κόστος. Επομένως, δεν ε, έχουμε ξεκινήσει ταυτόχρονα την έρευνα, όπως έχουμε με την περίπτωση του διαχειριστή δικτύου, γιατί μας είπαν οι γερμανικές αρχές ότι προετοιμάζουν ένα νομοθεσία. Και εγώ τους είπα, εντάξει, ας δούμε την νέα νομοθεσία και θα λάβουμε υπόψη το νέο καθεστώς, όχι μόνο το αρχικό πρέπει να λάβουμε κάποια απόφαση για το τι θα κάνουμε. Πρόσφατα ήμουν στο Βερολίνο και συζήτησα με τον Δικακελάριο και τον Υπουργό. και μας είπαν ότι τον Ιούνιο περίπου θα λάβουμε νέες πληροφορίες σχετικά με το νέο σύστημα. Αν όχι, θα αναγκαστούμε να ανοίξουμε έρευνα για την προηγούμενη περίπτωση. Για τη χαλιβουργία, ναι, απάντησα. Έβαλα και ένα αλλά στο τέλος βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ταξίζει να μένει κανεί μέχρι το τέλο, να υπενθυμίσω σε όλου, ότι σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας στις 3.30 στην Α53 αίθουσα και θα έχουμε την ακρόαση για τη ΦΑΤΚΑ, για το νόμο για την επιβολή φορολογία του λογαριασμού αλλοδαπής.